Thank you, Thank you, colleagues, uh, Ευχαριστώ συνάδελφοι και να καλωσορίσω καταρχήν τους εκπροσώπους από τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή πριν να αρχίσουμε με την ακρόασή μας. Το σημείο 1 της ε, ημερήσιας διάταξης αφορά ένα νέο σημείο 5.1 η παρουσίαση των ε, διαπραγματεύσεων τριμερές διάλογο για την καταπολέμηση της απάτης και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σημείο 5 για την ε, αποστολή στο Λίβανο 19-22 Σεπτεμβρίου θα γίνει αύριο στις 9. Και το θέμα των μεταναστευτικών ε, ε, ροών σε σχέση με την ΕΙΕΔ θα αναβληθεί. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη από γλωσσικής πλευράς. Δεν έχουμε κερτικά, ε, ε, ελληνικά, εσθονικά, τσεχικά και τα τσεχικά μάλλον θα είναι παθητική γλώσσα. Στα σημεία 3, στο σημείο 3 έχουμε εγκρίνει τα πρακτικά της 17ης Μαρτίου και του Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Καλωσορίζουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια και φυσικά τους δικούς μας Ευρωβουλευτές για αυτή την διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Εθνικών Κοινοβουλίων για την ε, υλοποίηση της Ένωσης Ασφάλειας και το ρόλο της Ευρωπόλ. Γνωρίζουμε πολύ καλά και ιδιαίτερα οι ευρωβουλευτές το γνωρίζουν ότι υπάρχει μια ειδική ατζέντα για την ασφάλεια της Ένωσης με βάση ακριβώς αυτή την ένωση όπως έχει διαμορφωθεί. Έχουμε το νέο Επίτροπο για θέματα ασφάλειας και φυσικά υπάρχει εποπτεία και έλεγχος και καλή εταιρική σχέση με την Europol, η οποία συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Κίνγκ και τον Διευθυντή της Ευρωπόλ. Θα συστήσουμε λοιπόν σήμερα ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την ε, ατζέντα της ασφάλειας και τι σημαίνει αυτό για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα θέλαμε να είναι μια ουσιώδης ε, συζήτηση και όχι διακοσμητικού χαρακτήρα. Χαίρομαι λοιπόν γιατί έχουμε 46 μέλη εθνικών κοινοβουλίων που προέρχονται από 23 κράτη-μέλη και μία χώρα του ΕΟΧ. Κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα εθνικά κοινοβούλια για τα θέματα ασφαλείας και ιδιαίτερο το ρόλο της ε, Europol. Θα ήθελα λοιπόν συνάδελφοι αμέσως να περάσουμε στην ε, πρώτη μας, ε, στο πρώτο μας πάνελ. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο και γνωρίζω ότι πολλοί θα θέλατε να λάβετε το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Γι' αυτό και περνάμε και στην πρώτη μας συνεδρίαση για το γενικό πλαίσιο, την υλοποίηση της Ένωσης Ασφάλειας και το ρόλο της ε, Ευρωπόλ στα πλαίσια αυτής της ασφάλειας για την ε, επιχειρησιακή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο της ε, Ευρωπόλ. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Τζούλιαν Κίνγκ και το Διευθυντή της ε, Ευρωπόλ. Θα ήθελα να πω ότι οι ερωταποκρίσεις βασίζονται σε έναν πολύ ε, δύσκολο ας πούμε προσδιορισμό χρόνου και εάν θεωρείτε ότι δεν ε, έχετε λάβει το λόγο να το αναφέρετε. Σε σχέση με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων θα θέλαμε με, αυτές τις, ε, με αυτά τα δελτία να αναγράψετε τα δελτία αυτά, να αναγράψετε το όνομά σας για να λάβετε το λόγο, για να γνωρίζουμε ότι θέλετε να λάβετε το λόγο. Και αν σας ξεχάσουμε να μας το αναφέρετε με ανάταση του χεριού ε, ως προς δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί τους αναγνωρίζω. Λοιπόν, θα θέλαμε ε, να ε, μας αναφέρετε με αυτά τα δελτία, με διανατάσεις ισχυρός, να μας πείτε αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Α, με συγχωρείτε, θα πρέπει επίσης να σας πω ότι υπάρχει και ο, ο Ντομινίκ Ράμπορκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Πράξεων νομοθεσίας και Γενικής Διοίκησης της Γαλλικής Συνέλευσης ο κύριος Ντομινίκ Κρεμπούρκ και χαίρομαι γιατί και οι τρεις ε, ομιλητές είναι μαζί μας. Αρχίζουμε λοιπόν με τον Επίτροπο Τζούλιαν Κίνγκ, ο οποίος ασχολείται με την Ένωση Ασφάλειας θα λάβει το λόγο για 10 λεπτά και θα μας πει πώς ακριβώς βλέπει την Ένωση Ασφάλειας να διαμορφώνεται και τον ρόλο του μέσα στα πλαίσια αυτή τη Ένωση Έχετε το λόγο. Διευκρίνησε την ελληνική καμπίνα υπάρχει διερμηνία και από και προ ελληνικά. Χαίρετε λέει ο κύριο Κέιν. Χαιρετίζω την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά <clears throat> και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η Επιτροπή φυσικά λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας λογοδοτώ απευθείας στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον πρόεδρο Γιούνκερ να αναπτύξει στενότερε σχέσει με τα εθνικά κοινοβούλια. Και στηρίζω πλήρω τι δεσμεύσει που έχει κάνει ο πρόεδρο Γιούνκερ από αυτού τι τελευταίε εβδομάδε. Είχα ανταλλαγή απόψεων με το Εστονικό Κοινοβούλιο, το Γερμανικό Bundestag, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το Ιταλικό Κοινοβούλιο και την Βρετανική Βουλή των Λόρδων. Και Προσβλέπω σε περαιτέρω τέτοιε ανταλλαγέ απόψεων στι προσεχείς εβδομάδε και μήνε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λογοδοτεί ακόμη περισσότερο στα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχουν ε, διαδικασίε διαμόρφωση πολιτική που μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικέ και διαφανεί εάν υποφελούνται από μια τέτοια στενή σχέση. Και η διαμόρφωση πολιτική υποφελείται ε, από τέτοιε σχέσει με τα εθνικά κοινοβούλια και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για την εργασία των οργανισμών της Ένωσης που παίζουν ζωτικό ρόλο για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Στην κοινή μας εργασία για μια Ένωση Ασφάλειας η Europol παίζει κεντρικό ρόλο για πολλές πολιτικές και πολλά μέσα που αποφασίζει η Ένωση. Ο νέος κανονισμός για την Europol που όπως ξέρετε θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Πέμπτη του 2017 θέτει νέες προδιαγραφές για κοινή, κοινό, δημοκρατικό έλεγχο και από το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες για ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο της Europol και για τον ε, κοινό έλεγχο μέσω του, της κοινή ομάδας κοινοβουλευτικού έλεγχου. Χαιρετίζω λοιπόν την συνεδρίασή μας σήμερα ως ένα πρώτο βήμα για να εφαρμοστεί αυτή η πρακτική κοινοβουλευτικής επιτήρησης. Δεν θα σας αναφέρω αναλυτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα περίπλοκο σύνολο από απειλές ασφαλείας πολύ σημαντική, τη σημαντικότερη για πολλά χρόνια τρομοκρατική απειλή. Ο συνάδελφος ε, και φίλος Ρομπ Wainwright θα σας πει λίγο περισσότερα για το πώς διαμορφώνεται αυτή η απειλή. Αλλά υπάρχει μια προφανής ευρωπαϊκή διάσταση. Ούτε η τρομοκρατία, ούτε το οργανωμένο έγκλημα σταματούν σε σύνορα. Αν εξετάσουμε τις πρόσφατες επιθέσεις, πολλές πλευρές της προετοιμασίας και εκτέλεσής τους ήταν διεθνικές. Οι τρομοκράτες, δυστυχώς, δεν ε, εστιάζουν στο α ή το β κράτος μέλος, στοχεύουν τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή διάσταση στην ε, αντίδρασή μας. Τις αντιδράσεις μας λοιπόν στην τρομοκρατία, στο κύβερνο έγκλημα και την κύβερνο απειλή και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό είναι ένας από τους λόγους επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση του Πρόεδρου Γιούνκερ το περασμένο καλοκαίρι να υπάρξει ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για την ε, Ένωση Ασφάλειας. Όλα αυτά βεβαίως έχουν στο επίκεντρό τους την Europol. Η, Ένωση, η Europol παίζει ουσιώδη ρόλο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές. Και θέλω να χαιρετήσω τη θαυμάσια εργασία που έχει κάνει ο Ρομπ και όλους τους αφοσιωμένους συνεργάτες του στη Europol, άνδρες και γυναίκες. Έχουν ε, μοναδικές δυνατότητες καταπολέμησης του εγκλήματος, έχουν ένα σύστημα πανευρωπαϊκό ανταλλαγής πληροφοριών, κάνουν καταπληκτικές αναλύσεις, έχουν ρωμαλαίο σύστημα προστασίας των δεδομένων. Η ανάλυση των απειλών που έχουν κάνει, σε συνεργασία με τις ε, αστυνομικές αρχές σε όλες ε, τις χώρες μέλη, μας καθορίζουν, μας βοηθούν να καθορίσουμε τους κοινούς μας στόχους και ακόμη και πριν το νέο κανονισμό της Europol, η Europol είχε δομηθεί με βάση την αντιπολέμηση αυτών των απειλών. Τρομοκρατία, κυβερνοέγκλημα, οργανωμένο έγκλημα. Το κέντρο που έχει, ε, ε, έχει δημιουργήσει η Europol μας βοηθάει να καταπολέσουμε την τρομοκρατία. Είναι ένα κέντρο Ανταλλαγή πληροφοριών, μα ε, βοηθάει να, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της χρηματοδότηση, της τρομοκρατίας, της επιγραμμικής προπαγάνδας, του παράνομου εμπορίου, του λαθρεμπορίου όπλων και των ε, ξένων μαχητών. Και αυτό το κέντρο έχει ήδη αποδείξει την αξία της γιατί δίνει βοήθεια στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τι φρικτέ τρομοκρατικέ απειλέ που υπήρξαν νωρίτερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Το κέντρο εγκλήματος είναι πόλος που δίνει βοήθεια και συντονίζει εκατοντάδες επιχειρήσεις. Συλλέγει και διανέμει στοιχεία για χιλιάδες εγκληματίες και δημιούργησε νέα αποτελεσματική συνεργασία, εντοπίζει εγκληματίες και καταφέραμε να διασώσουμε χιλιάδες παιδιά από κακοποίηση μέσω του ίντερνετ. Επίσης, Έχουμε και το κέντρο κατά του λαθρεμπορίου που βοηθάει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα δίκτυα λαθρεμπορίου και η Europol συμβάλλει στον κύκλο πολιτική της Ένωσης για το οργανωμένο σοβαρό διεθνές έγκλημα. Η αποτίμηση των εγκληματιών βοηθάει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν προτεραιότητες και κοινέ δράσεις. Η Επιτροπή στηρίζει τι σημαντικέ αυτέ πτυχέ τη Europol και των κέντρων της παρέχοντας τους πόρους που απαιτούνται και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του. Φέτος το Europol πήρε 36 νέες θέσεις και τώρα έχει σχεδόν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των σκελών της αρχής του προπολογισμού για άλλες 60 θέσεις στον προπολογισμό του 17 και η Κομισιόν και το Europol ξεκινήσανε μία αποτίμηση των αναγκών για να δουν τι μελλοντικέ ανάγκες θα είχαμε. Λόγω όλης αυτής της εργασίας η Europol πρέπει να θεωρούμε ότι δικαιολογεί την ύπαρξή τη ε, στην κοινή γνώμη. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια μπορεί να γίνει μόνο πραγματική και βιώσιμη όταν οι πολίτε είναι πεπισμένοι, έχουν εμπιστοσύνη ότι γίνονται απολύτω σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Ακόμη και υπό του παλαιότερου κανόνε, η Europol είχε ένα ρωμαλαίο πλαίσιο προστασία των δεδομένων. Ορισμένοι λένε το πιο ρωμαλαίο, το πιο έντονο πουθενά στον κόσμο. Και αυτό έχει έννοια. Οι εθνικές αρχές αστυνόμευσης πρέπει να είναι σίγουρες ότι οι πληροφορίες ε, που μοιράζονται με την Europol προστατεύονται από την Europol. Το νέο πλαίσιο τώρα εξυγχρονίζει και περαιτέρω ενισχύει αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει σημαντικό ρόλο για τον επιτηρητή προστασία των δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτηρεί τη διαδικασία επεξεργασία των δεδομένων από την Europol. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η συζήτησή μα σήμερα, η ομάδα κοινού κοινοβουλευτικού ελέγχου θα αυξήσει περισσότερο την διαφάνεια και λογοδοσία της Europol. Θα ενισχύσει έτσι την νομιμοποίησή της. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στη δημιουργία αυτών των διαδικασιών για να ε, παίξει το ρόλο του ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με βάση τους ρόλους που καθορίζει ο νέος κανονισμός. Η Europol είναι οργανισμός κλειδί και η συμμετοχή σας οπωσδήποτε θα την ενισχύσει περτέρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Όπω είπε ο Επίτροπος, ο νέο κανονισμό Europol θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαου του 2017. Στην επόμενη ενότητα οι ευρωβουλευτέ θα εξετάσουν πιο συγκεκριμένα ε, τη συμφωνία για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτό το έχετε εξετάσει σε μεγάλο βαθμό και στα εθνικά κοινοβούλια. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον ε, διευθυντή τη Europol, για να μας ε, μιλήσει πώς ακριβώς εντάσσεται η Europol αυτή τη στιγμή στις ευρύτερες εξελίξεις ε, της ασφάλειας, της, της Ένωσης Ασφάλειας και όπως ανέφερε προηγουμένως ε, και ο κύριος Κιν, να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Έμγρατ για την συνεργασία της Europol μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την συνεχή στήριξή τη ε, και μεμονωμένα από επιμέρου ευρωβουλευτέ, αλλά και συνολικά για τη στήριξη σα, λοιπόν ιδίω ό,τι αφορά την ε, ολοκλήρωση ε, του νέου κανονισμού Europol και για τη στήριξη και του Επιτρόπου κ. Κίνγκ αλλά και για των μελών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που μας έδωσαν και περισσότερους πόρους. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για την στήριξη που λάβαμε και από πολλά εθνικά κοινοβούλια, όπω ανέφερε και ο κύριο ε, Επίτροπο ε, του τελευταίου μήνε και έτη. Ευχαριστώ πολύ. Προ τον ε, κύριο Επίτροπο, λοιπόν, μα έχει στηρίξει πάρα πολύ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και μας έχει βοηθήσει στη Europol να αναπτύξουμε τις δυνατότητές μας σε ό,τι αφορά νέες, πιο σύνθετες και πολυδιάστατε προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα ήθελα να σταθώ μερικά λεπτά για το πώς ακριβώς η Europol ε, πρακτικά ε, ωφελεί και βοηθά τα κράτη-μέλη ενώπιον αυτών των απειλών. Ξέρετε ότι η Europol δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό FBI. Ανταυτού βοηθούμε τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία με, την, με το να τους παρέχουμε τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, ιδίως σε ό,τι αφορά το, την κρίσιμη σημασία ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε ένα μοναδικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με πάνω από 750 ε, αρχές ε, ανά την Ευρώπη και άλλες ε, χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά, όπως είναι η ΙΠΑ, η Ελβετία και η Νορβηγία μια πολύ μεγάλη διασυνδεδεμένη κοινότητα ε, των αρχών επιβολή του νόμου που ανταλλάζει χιλιάδε πληροφοριών κάθε μέρα σε ό,τι αφορά το σοβαρό έγκλημα και τι δημοκρατικέ οργανώσει. Και αξιοποιούμε αυτή την αναλυτική μας ικανότητα ε, και έτσι μπορούμε ε, να εντοπίσουμε την διασυνοριακή δραστηριότητα και έτσι να δώσουμε στις εθνικές αρχές αυτά που χρειάζονται για να ε, διενεργήσουν ε, τις αστυνομικές και άλλες ε, επιχειρήσεις τους και δραστηριότητες για να σταματήσουμε τις επιθέσεις αυτές και γενικά αυτές τις εγκληματικές ενέργειες που μας πλήττουν. Έχουμε μερικούς από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη για το κυβερνοέγκλημα, την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο κτλ. Έχουμε 200 ε, επιτετραμένους ε, που συνδράμουν σε αυτήν την διαδικασία και χρησιμοποιώντας τη δική μας προγνωμοσύνη μπορούν να συντονίζουν ε, διασυνοριακές επιχειρήσεις μέχρι και 40.000 υποθέσεις ανά χρόνο έχουμε που περνάνε μέσα από τα χέρια της Europol. Για παράδειγμα, ε, θα αναφέρουμε την επιτυχή ολοκλήρωση ε, και διάλυση ενός ε, εγκληματικού δικτύου στην Ισπανία. Επίσης, έχουμε κατεβάσει πάνω από 4.500 παράνομους ιστοτόπους που αφορούσαν το λαθρεμπόριο παραποιημένων προϊόντων. Υπάρχει λοιπόν μία συνεχή δραστηριότητα για να δώσουμε προσθεμένη αξία στις ε, δράσεις των κρατών μελών για την καταπολέμηση του, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου κυβερνού Αν δείτε και τα στατιστικά στοιχεία, έχουμε εξαπλάσιες πληροφορίες ε, πλέον που επεξεργάζεται η Europol αυτή τη στιγμή σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια και τετραπλάσιος αριθμός υποθέσεων στον οποίο ε, παρέχει τη στήριξή της ε, η Europol. Αυτό δείχνει πως έχει εξελιχθεί η ευρύτερη εικόνα ε, του κυβερνοεγκλήματος και της τρομοκρατίας ακόμα και μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια. Είναι πλέον πιο παγκοσμιοποιημένη υπερεθνική διεθνική διαργασία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε την Ένωση Ασφάλειας. Βλέπουμε και μέσω των τρομοκρατικών επιθέσεων ποια είναι η κλίμακα πλέον ε, στην Ευρώπη από τον αριθμό των επιθέσεων, τον αριθμό των θυμάτων, τον αριθμό των αλλοδαπών μαχητών που από τις δικές μας κοινότητες έχουν μεταβεί ε, στη Συρία και στο Ιράκ. Ξέρουμε ότι, ή εκτιμούμε ότι περίπου 5.000 έχουν επιστρέψει ε, στην Ευρώπη και αποτελούν επιλή για τις κοινωνίες μας. Βλέπουμε πόσο σύνθετη είναι αυτή η εικόνα, γιατί έχουμε και πολλούς ε, μοναχικούς λύκους που από τα σπίτια τους, ενώ είναι μόνοι, χωρίς κάποια άλλη διασύνδεση, λαμβάνουν αυτή την έμπνευση να διενεργήσουν αυτές τις ε, φρικτές επιθέσεις. Χρήση τεχνολογίας, ό,τι φορά την διάδοση αυτής της άσχημης ρητορικής που αξιοποιεί ο ISIS με έναν τρόπο πρωτοφανή. Έχουν αλλάξει λοιπόν πολύ τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία. Γι' αυτό και για πρώτη φορά, όπω είπε και ο Επίτροπο Κίνγκ, ε, έχουμε ένα ευρωπαϊκό ε, κέντρο αντιτρομοκρατία που μπορεί να βοηθήσει στα κράτη-μέλη σε αυτή τη κρίσιμη σημασία συνταλλαγή πληροφοριών και την ε, διασύνδεση των δύο τομέων του κυβερνοεγκλήματο και τη τρομοκρατία. Το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό Έχουμε μια ειδική μονάδα που βοηθά τις αστυνομικέ αρχές ανά την Ευρώπη ε, να εξετάζουν τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων για να εντοπίζουν ε, τρομοκρατική προπαγάνδα και να την αφαιρούν από το διαδίκτυο. Υπάρχει κεντρικό σημείο επαφής. Η μονάδα μας λοιπόν συνεργάζεται με 60 τέτοιες ε, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αφαιρεί χιλιάδες τέτοιους λογαριασμούς και μηνύματα κάθε χρόνο παρακολουθούμε χρηματοδοτικές ροές ε, της τρομοκρατίας και παρέχουμε και σημαντική επιχειρησιακή αρρωγή σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση πιο συγκεκριμένα των επιθέσεων σε Βρυξέλλες και Παρίσι ε, για τον αντοπισμό των ε, υπολείπων μελών αυτών των δικτύων και θέλουμε και μάλλον βοηθούμε για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον οι εγκληματικές ομάδες προσπαθούν να αξιοποιήσουν ε, ε, την προσφυγική κρίση. Αυτό συνέβη ιδίω το 2015 μέσω ε, την εμπορία ανθρώπων και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσπαθούσαν λοιπόν να εκμεταλλευτούν τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, των προσφύγων που προσπαθούσαν να μπουν στην Ευρώπη και το 2015 και έως και σήμερα. Έως 90% όλων των αφιχθέντων στην Ευρώπη το 2015 έλαβαν διευκόλυνση σε τουλάχιστον ένα τμήμα του ταξιδιού τους από τέτοιες ε, εγκληματικές ε, οργανώσεις. Θεωρούμε ότι ε, η εμπορία ανθρώπων θα πρέπει να τεθεί, οι διακινητές δηλαδή, θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος γιατί συνδέεται και με τα δύο ζητήματα. Έχουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, διακίνηση Ανθρώπων που έχει εντοπίσει πάνω από 50.000 ε, διακινητές που θεωρούμε ότι συμμετέχουν ε, σε, στην εμπορία ανθρώπων σήμερα στην Ευρώπη. Παρακολουθούμε πώς Αυτέ οι εγκληματικέ δραστηριότητε συνδέονται με άλλε μορφέ εγκληματική δραστηριότητα. Μα απασχολεί ο αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων, των παιδιών δηλαδή που έρχονται ε, με το προσφυγικό κύμα και πώ κάποιοι από αυτού τουλάχιστον μπορούν ε, να πέσουν θύματα εκμετάλλευση από αυτέ τι εγκληματικέ οργανώσει. Και οποιαδήποτε προσπάθεια ε, των ε, τρομοκρατικών ε, οργανώσεων σίγουρα θα περιλαμβάνει και μια τέτοια κίνηση και στοχοθέτηση του προσφυγικού κύματος. Το κυβερνοέγκλημα είναι εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα στοιχεία γιατί είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο σήμερα διευκολύνει το έγκλημα και εδώ είναι τεράστια η κλίμακα και αυξάνεται εκθετικά σε ό,τι αφορά την, ε, ε, συγγνώμη, τις ε, επιθέσεις στο διαδίκτυο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφεσε θύμα μιας τέτοιας επίθεσης των ΧΑΚΕ την περασμένη εβδομάδα. Έχει εξαπλασιαστεί λοιπόν ο αριθμός αυτών των επιθέσεων μέσα σε ένα χρόνο. Πολλές φορές έχουμε, ε, ζητούνται λίτρα και πλέον έχει γίνει ο καταξεχήν τρόπος επίθεσης στο διαδίκτυο και στο, Τοχοποιούνται πλέον ακόμα και νοσοκομεία και ε, άλλοι φορείς. Βλέπουμε το εύρος και τις δυνατότητες που υπάρχουν για ε, την ε, κακοποίηση και σεξουαλική και εκμετάλλευση ανηλίκων τα τελευταία χρόνια. Και αυτό γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση πλέον μέσω του διαδικτύου. Έχουμε και το ίντερνετ, το διαδίκτυο των αντικειμένων, το οποίο έχει αυξήσει τις δυνατότητες για τους εγκληματίες και βλέπουμε ε, μια δυναμική δημιουργίας ε, όλο και πιο διασυνδεδεμένων ε, συσκευών και τεχνολογιών, αλλά χωρίς να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τους κινδύνους που δημιουργούνται, ιδίως προς τους ανηλίκους, που είναι πιο ευάλωτοι. Το 2013 διαμορφώσαμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή παρέχει στήριξη σε 200 ε, υποθέσεις ε, υψηλού προφίλ κάθε χρόνο. Έχουμε και καινοτόμες ε, εκστρατείες όπως είναι η εκστρατεία για το τερματισμό της παροχής λίτρων δίνει μια δωρεάν υπηρεσία ε, αποκρυπτογράφηση στα θύματα τέτοιων επιθέσεων με λίτρα και είχαμε 15 εκατομμύρια επισκέπτες ε, στον ιστότοπο και μεγάλο αριθμό ε, ανθρώπων που κατέβασαν αυτό το δωρεάν λογισμικό από κρυπτογράφησης ή από κωδικοποίησης. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο περιβάλλον πιο σύνθετο, πιο διασυνδεμένο. Γι' αυτό και η δική μας ανταπόκριση θα πρέπει ε, να κινηθεί ε, σε, σε ένα γνώμονα ισχυρών και διασυνδεμένων δικτύων. Και η Europol αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Αρχών Επιβολής του Νόμου ε, να λαμβάνει την αρρωγή της Europol. Βλέπουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τα δεδομένα για να έχουμε μια καλύτερη απάντηση ενώπιον αυτών των απειλών. Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα νέο σύγχρονο καινοτόμο τρόπο για την καταπολέμηση των νέων διασυνοριακών ε, απειλών ασφάλειας. Ο κόσμος μας λοιπόν γίνεται πιο σύνθετο και σημαντικό τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας είναι ότι ε, τα ε, επίπεδα λογοδοσίας μας θα πρέπει να παραμείνουν ιδιαίτερω υψηλά. Λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήδη έχουμε ιδιαίτερα εύρωστα μέτρα σε ό,τι αφορά την ε, προστασία δεδομένων, ιδίω εφόσον υπάρχει και συστηματικός έλεγχος ε, από το ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς λογοδοτούμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως ε, λέει και ο Πρόεδρος και εγώ προσωπικά αλλά και ε, ο φορέας μου όλο ένα και περισσότερο θα λογοδοτούμε ε, σε εσά και στα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό το στηρίζουμε εμεί ω φορέα για να αυξήσουμε τη δημοκρατική μα νομιμοποίηση και την αξιοπιστία ε, στα μάτια του, των πολιτών. Γι' αυτό θέλαμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν την ε, κοινή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου και προβλέπουμε σε συνέχεια την εργασία μα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε αυτά τα θέματα ελέγχου και στην επόμενη συνεδρία μας. Και τώρα θα δούμε την ε, προοπτική από τον εκπρόσωπο μιας χώρας που έχει πληγεί από θέματα ασφάλειας από τον Ντομινίκ Ρεμπούρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Πράξεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Κυρίε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι η μαρτυρία από έναν κοινοβουλευτικό ε, εκπρόσωπο μιας χώρας που έχει ιδιαίτερα πληγή είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι η Γαλλία έχει πληγεί ιδιαίτερα και 240 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και το Βέλγιο έχει πληγεί και θα ήθελα να αποτίσω ένα φόρο τιμής σε όλα αυτά τα θύματα και σε όλους εκείνους οι οποίοι τραυματίστηκαν και ακροτηριάστηκαν. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η διεθνής συνεργασία είναι ύψης της σημασίας. Αυτό είναι αυτονόητο και το είπατε κι εσείς κύριε Επίτροπε. Η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα έχει διεθνικό χαρακτήρα και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκές λύσεις σύμφωνα με τις αξίες της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω τη δημιουργία της συνοριοφυλακής που έγινε μέσα σε ένα χρόνο ενώ την περιμέναμε εδώ και δέκα χρόνια καθώς και το το PNR το οποίο ε, ολοκληρώθηκε καθώς και τον διορισμό ενός επιτρόπου για θέματα ασφαλείας, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι η οδηγία κατά της τρομοκρατίας που συντάσσεται τώρα θα επιτρέψει την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών μέσα στα πλαίσια των στρατιωτικών επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες που χρειαζόμαστε άμεσα. Θα ήθελα να επιτελεστεί πρόοδος σε πολλές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα και ξέρουμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διάδοσή τους πέρα από τις αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Επίσης, ε, όπως ε, είπατε πολύ σωστά, έχει μεγάλη σημασία η καταπολέμηση και η ποινική δίωξη των ε, υπετίων και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα Μητρώα και ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο επ' αυτού. Και φυσικά η παρέμβαση του προσωπικού στα hot spots. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών αρχών και εθνικών κοινοβουλίων και επειδή οι αστυνομικές δραστηριότητες θα πρέπει να διοργανώνονται μέσα στα πλαίσια ενός ελέγχου και εποπτείας αυτών των δραστηριοτήτων. Γι' αυτό υπάρχει και η Μικτή Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που θα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα αλλά που θα συμμετάσχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή Προεδρία, Ευρωπαϊκή και εθνική μέσα στα πλαίσια των εκπροσώπων που προσέρχονται συχνά και ασχολούνται από αυτό το ζήτημα. Δεν ε, είμαι ωφελημιστής και δεν έχω ιστερόβουλες σκέψεις, γιατί ξέρετε ότι η δική μου θητεία λύγει πολύ σύντομα. Εν πάση περιπτώσει μίλησα για μια αναγκαιότητα και νομίζω ότι και εθνικοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Ντομινίκ. Φυσικά, ένας πολιτικός πάντα θα πρέπει να έχει κίνητρα. Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα θα ε, λάβουν το λόγο δύο εκπρόσωποι από εθνικά κοινοβούλια και στη συνέχεια ένας ευρωβουλευτής. Έτσι θα συνεχίσουμε και με αυτό το ε, διάλογο με βάση τη σειρά δήλωσης. Να μου πείτε αν δεν ακούσετε το όνομά σας. Από τα Εθνικά Κοινοβούλια λοιπόν Κυρία Καρμαλή έχει το λόγο. Είναι αντιπρόεδρος υπεύθυνη για θέματα ε, ευρωπαϊκής ασφάλειας και κοινωνικών υποθέσεων και εκπροσωπεί την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Συνάδελφοι, θα ήθελα να περιοριστείτε στα δύο λεπτά σας παρακαλώ. Να παρακολουθείτε και το ρολόι σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους παρεμβαίνοντες. Μιλήσατε για σημαντικά διακυβέρματα σήμερα ως προς την Ευρωπόλ και γενικότερα θέματα ασφάλειας. Θα ήθελα να αρχίσω με την έκθεση του Μαρτίου του 2016 του Ευρωπαίου Συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εκεί βλέπουμε ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος, αλλά πολλά υπολείπονται, γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε. Ιδιαίτερα για την Ευρωπόλ, τα προσωπικά δεδομένα, την έκθεση Προύμ, το PNR όπως προείπα, και θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. 1.500 άτομα που ορίστηκαν βρίσκονταν στο Μητρό της Ευρωπόλ που μετέβησαν στο Ιράκ και στη Συρία για να προσχωρήσουν στη ΝΤΑΕΣ, αλλά ο συνολικός αριθμός είναι 5.000. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μεγάλη συνεργασία και κοινή διαχείριση. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα κατάλληλα μέσα για να εφαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή από πλευρά κονδυλίων και ουσίας γενικότερα για να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία. Προσκρούμε σε δυσκολίες, το ξέρουμε αυτό. Ελέγχθη πολλές φορές και ως προς το διαλειτουργικό πλαίσιο. Πρόκειται για τεχνικής υφής δυσκολίες ή υπάρχουν πολιτικές αμφιβολίες σε σχέση με ένα νέο πεδίο δράσης το οποίο ήταν πολύ περιορισμένο, πολύ συσταλτικό πριν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μία πορεία, μία χαρτογράφηση καθώς και χρονοδιάγραμμα για αυτά τα μέσα που είναι ευρωπαϊκού και εθνικού χαρακτήρα. Ως προς το θέμα της Ευρωπόλ και του κανονισμού της, κατά τις ακροάσεις στην Γαλλική ε, Εθνοσυνέλευση και τις προτάσεις νόμου, είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ανεπάρκειες σε σχέση με τον κανονισμό της Ευρωπόλ και ιδιαίτερα για την προστασία δεδομένων. Και για τη συμφωνία ενός ε, κράτους μέλους για να μεταφερθούν ε, αυτά τα δεδομένα και αυτό αφορά και τρίτες χώρες για την διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες, κάτι το οποίο ε, επιβάλλει προγενέστερη ε, απόφαση και αδειοδότηση και αυτό μέσα στα πλαίσια ενός έτους. Θα ήθελα μία απάντηση κατά το δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας υπενθυμίσω, συνάδελφοι, ότι είναι πραγματικά τα δύο λεπτά, όχι εικονικά. Θα ήθελα να βλέπετε το, το ρολόι το οποίο σας χρονομετρεί για να έχουμε ώρα και για απαντήσεις. Lord Sally. Από την, ε, την ε, Γερουσία, από το House of Lords, όποια και να είναι η απόφαση ενδεχόμενης απαχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν την στενότερη δυνατή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Ξέρω από πικρά πείρα ότι είναι πολύ δύσκολο να εξισορροπήσουμε τις πολιτικές ελευθερίες τις οποίες υπερασπιζόμαστε με την ασφάλεια. Ασφάλεια προς τους πολίτες και όταν γίνεται μία τρομοκρατική ενέργεια πολλοί ζητούν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, αλλά όταν γίνει κακή χρήση προσωπικών δεδομένων, τότε θα πρέπει να γίνει μια συσταλτική ερμηνεία της ασφάλειας. Γι' αυτό νομίζω ότι και στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό βεβαίως έχουν έναν κρίσιμο ρόλο για αυτή την εξισορρόπηση μεταξύ πολιτικών ελευθεριών και ασφάλειας των πολιτών. Χρειάζεται συνεχής εποπτεία που μπορεί να γίνει μόνο από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εμείς προσχωρήσαμε στην Ευρωπόλ πρόσφατα και ελπίζω να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας στο τομέα της ασφάλειας, γιατί αυτό ακριβώς δεχτήκαμε και θα πρέπει να το υλοποιήσουμε και νομίζω ότι όλα αυτά τα είπα μέσα σε δύο λεπτά. Ναι, ναι, εξοικονομήσαμε και 15 δεύτερα. Τώρα από τους ευρωβουλευτές, ο κύριος Δίας Τεμέρα ε, έχει το λόγο. Ήταν ε, εισηγητής για θέματα Ευρωπόλ ε, εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος προέρχεται από την Ισπανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαιρετίζω όλους τους συζητητές μας ε, σε αυτό το γύρο συζητήσεων. Θέλω να παρέμβω για λόγους ευγένειας και να κάνω μια διευκρίνηση. Η διευκρίνηση που θέλω να κάνω είναι, είναι ότι η Europol είναι ένα αναγκαίο μέσο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα βοηθήσουμε αυτό το φορέα και ο φορέας ε, ε, χέρι της πύρους εμπιστοσύνης μας. Δεύτερον, μια διευκρίνηση προς τη Γαλλίδα συνάδελφα που μόλις παρνεύει. Όχι, δεν είναι σχέδιο κανονισμού αυτό που έχουμε ενώπιον μας. Είναι ένας κανονισμός, ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία στις 11 Μαΐου τρέχοντος. Λοιπόν, η νομική προσωπικότητα της Europol θα αρχίσει να λειτουργεί από τον επόμενο Μάιο. Δεν χρειάζεται μεταγραφή στην εθνική νομοθεσία. Δεν πρόκειται για οδηγία. Ένας κανονισμός από την 1η Μαΐου, όπως κάθε κανονισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σεβαστός από τα κράτη-μέλη. Το σύστημα της προστασίας δεδομένων που σας απασχολεί είναι ιδιαίτερα ρωμαλαίο, όπως είπε ο Επίτροπος. Και υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι με τους οποίους το συζητάω, όπως ο Μόρτεν Πέτερσεν, είναι ο Τέρι Κάμπρας, ο Ιωζέπ και άλλοι από διάφορες πολιτικές ομάδες. Όλοι αυτοί συνεργάστηκαν μαζί μου για την εκπόνηση αυτού του κανονισμού. Και είναι λοιπόν ένα μέσο, ένα ουσιώδες, θεμελιώδες εργαλείο. Όλα όσα υπόθηκαν θα υπογραμμίζω όλα τα κέντρα και για κάτι που δεν αναφέρθηκε για ε, λόγους ε, συντομίας, ο Οργανισμός για την Προστασία του Ευρώ. Και επίσης, ε, δεν θα αναφερθώ τώρα στην ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου γιατί θα τη συζητήσουμε μετά. Αλλά αυτό που θέλω να πω και φυσικά στηρίζω τις εργασίες της Τρόικα, όπως ακριβώς τις καθόρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω λοιπόν να πω ότι όταν θα αρχίσει να ισχύει αυτή η κοινή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Europol θα αποκτήσει πολύ περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση και αξιοπιστία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διαθντεμέρα. Ο κύριος Χερβόνεν Φόλκ από την Επιτροπή Δικαιοσύνης του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Α, με συγχωρείτε. θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών ε, αστυνομικών αρχών και συνεργασία με τη Europol. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι όντως πολύ ουσιαστικό τμήμα της εργασίας μας. Και τώρα που έχουμε ενώπιον μας και το Brexit και το γεγονός ότι η Ευρώπη ε, αφισβητείται από ορισμένου ω ε, το σωστό πλαίσιο για τη συνεργασία των κρατών μελών μα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση των μορφών τη ευρωπαϊκή συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να το τονίσουμε αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να συνεργαζόμεθα εμεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια και, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να ασκείται ο σωστός κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των εργασιών της Europol από κοινού. Είναι σημαντικό να είναι ουσιώδης αυτός ο έλεγχος, να είναι απλός, συγκεκριμένος και ταχύς. Αυτά είναι τα αποφασιστικά. Ούτως ώστε οι πολίτες να αναγνωρίζουν, να αισθάνονται ότι οι περιορισμένοι μας πόροι, οι κοινοί, αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Και επίσης χαιρετίζω το ότι ε, η Europol εργάζεται με βάση προτεραιότητες. Η Σουηδία θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό στους τομείς αυτούς όπου υπάρχει συνεργασία να υπάρχει σαφής καθορισμός των προτεραιότητων ε, διαμεθοριακό οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία και κυβερνοεγκληματικότητα. Από την Κύπρο ο κύριο Δημήτρη Δημητρίου, μόνιμη Επιτροπή, τη κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, Νομικών Θεμάτων. Των ενδιαφέρον τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Κυπριακή Δημοκρατία, να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται στο θεματολόγιο για την ασφάλεια και την ενίσχυση του ρόλου τη Europol. Οι έντονε ανησυχίε των πολιτών μα σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια αντανακλούνται στην άσκηση του δικαιώματο τη ψήφου τροφοδοτώντα μια σημαντική στροφή στην πολιτική σκηνή, όπω καθιερώθηκε στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ενίσχυση του ρόλου του Europol, ώστε να συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση των θετικών ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ορατότητα του θετικού αντίκτυπου τη Ένωση στου πολίτε τη Ευρώπη σε αυτή την περίοδο έντονου ευρωσκεπτικισμού. Φυσικά, Υπάρχει μια σειρά από βασικέ προκλήσει που αφορούν στην Europol, για τι οποίε θα πρέπει άμεσα να βρεθούν λύσει, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ενισχυμένο ρόλο στα πλαίσια τη Ένωση Ασφάλεια. Για παράδειγμα, το θέμα του Brexit και πώ μπορούν να μετριαστούν επιπτώσει από την έξοδο τη Βρετανία, ε, πώ θα εξελιχθεί η συμμετοχή τη Δανία στην Europol μετά το αποτέλεσμα του σχετικού δημοψηφίσματο, ακόμη πώ θα ενισχυθεί η συνεργασία με τον Frontex και άλλα σώματα και παράλληλα πώς θα αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη. Όσον αφορά στο ζήτημα τη ανάγκη για ενισχυμένη επιχειρησιακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, είναι φανερό ότι αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα τη επιτυχία τη Ένωση Ασφάλεια. Η Κύπρο, αν και δεν συμμετέχει στον χώρο του Σέγγεν και δεν αντιμετωπίζει στο παρόν στάδιο το μέγεθο του προβλήματο που υφίστανται άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τρομοκρατικέ επιθέσει, διαρευνά τρόπου συμμετοχή στον ρόλο στο κοινό σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών Σέγγεν 2. Επιπλέον, στα πλαίσια των προσπαθειών για συμβολή στον περιορισμό τη πρόσβαση τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων εγκληματικών δικτύων σε πηγέ χρηματοδότηση, που αποτελεί και προτεραιότητα στο πλαίσιο τη Ένωση Ασφάλεια. Η Κύπρο έχει συνάψει συνεργασία με την Europol σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών για το ζήτημα τη καταπολέμηση στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκόμες, παρακαλώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δύο λεπτά. Κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να βοηθάει ε, τα κράτη-μέλη που ε, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να επενδύσουν ε, στην ε, κυβερνοασφάλεια. Υπήρξε αυτή η αναφορά για το, στο κυβερνοέγκλημα και για τα όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα για την, την επίθεση, δηλαδή δεν μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο παραπάνω. Και σε ό,τι αφορά την Διερευνητική Επιτροπή για τα έγγραφα Παναμά, ακούσαμε πρόσφατος μία ενημέρωση από την Europol ότι ουσιαστικά είχαν ταυτοποιηθεί σύνδεσμοι με τη χρηματοδότηση τρομοκρατία, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, που συνδέεται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ε, σε ό,τι αφορά τα έγγραφα Παναμά και αυτό συνδέεται με πολλά κράτη-μέλη. Αυτά τα κράτη-μέλη ζήτησαν τη βοήθεια της Europol για να εντοπιστούν ακριβώς αυτά τα δίκτυα. Επίσης, ε, αναφερθήκατε την εμπορία ανθρώπων και πώς αυτό συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Όμως μήπω και εμεί κάνουμε ακριβώ το ίδιο, διευκολύνουμε την τρομοκρατία και την εμπορία ανθρώπων με το να μην προβλέπουμε ασφαλείς και νόμιμες ε, διόδου ε, πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κύριε Βέινμπρουκ, θα ήθελα να μας πείτε κάτι ακόμα για την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό λόμπι και άσκηση πιέσεων κατά των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να μας πείτε αν είναι απαραίτητη αυτή η πρόταση. Αναφερθήκατε στο PNR, όμως η πρόταση αυτή δεν καλύπτει τις ιδιωτικές πτήσεις. Είστε βέβαιος ότι καλύπτεται όλες τις πτήσεις που προσγειώνονται στην ε, νίκια του Λούζη κτλ για παράδειγμα, ένας ε, Σαουδάραβας πρίγκιπας, όπως αυτός που ε, πέρυσι συνελήφθη με εμπόρευμα ναρκωτικών ουσιών ουσίες από αυτές που καταναλώνουν συνήθως οι μαχητές του Άισις. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι δεν μπορούν να προσγειωθούν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια ε, τέτοιου είδους αεροσκάφη παρά το PNR. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάρι Χέντριξεν από την Διαρκή Επιτροπή Δικαιοσύνης της Νορβηγίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο θεωρώ ότι είναι όντω ε, ε, σημαντικό θεμελιώδη στοιχείο οποιασδήποτε ε, εύρυθμα λειτουργούσα ε, δικαιοσύνη και δημοκρατία, συγγνώμη, και είναι πολύ σημαντική σημερινή συνάντηση. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολλέ τέτοιε εκδηλώσει και πρωτοβουλίε ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Νορβηγικό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε τέτοιε διαδικασίε σε ό,τι αφορά την κοινή ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρόμαστε που τα χρονικά διαστήματα μα προσκαλείτε και σε άλλου ε, φορεί κοινοβουλευτική συνεργασία. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να υπενθυμίσω ότι η Νορβηγία και στο κάτω το παρελθόν έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον τη να ε, συμμετάσχει στο, στη νέα ομάδα κοινού κοινοβουλευτικού ελέγχου που διαμορφώνεται για την Europol. Η Νορβηγία έχει επιχειρησιακή συμφωνία με την Europol αλλά και με την ε, ΣΥΠΟΛ και τη Eurojust ε, και έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Εξαιτία και αυτή τη βούλησή μα, αλλά και τη γεωργική μα ε, θέση και συμμετοχή στην ενιαία αγορά, η νέα ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι κάτι το οποίο μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα θα ήταν αμοιβαία αποφελέ, θεωρώ αν ε, θα μπορούσε να ε, συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα κοινοβουλευτικού ε, ελέγχου η Νορβηγία. Επομένω, κατά τη συζήτηση και αναθεώρηση των κανονισμών αυτή τη νέα ομάδα, ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να διασφαλίσουν τη συμμετοχή και παρατηρητών από τι χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Συναδελφοί, θα κλείσει ο κατάλογος ομιλητών αυτή τη στιγμή, επομένω ε, δεν θα πάρουμε άλλες συμμετοχές. Είναι μακρύς ο κατάλογος ομιλητών και θέλουμε να ακούσουμε απαντήσεις ε, και από το πάνελ. Η κυρία Κοζόμπολη από την Ελλάδα. Κυρία Κοζόμπολη. Ε, ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ αφιερώνει ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο μέρος στο ζήτημα του ελέγχου της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό, μέσω των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Η διακοινοβουλευτική διάσκεψη θα συμμετέχει, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία ελέγχου, καθώς ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων θα εμφανίζεται ενώπιόν της σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2, 2β τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Θα με ενδιαφέρει να γνωρίζω τις απόψεις σας για το πώς θα μπορούσε η διαδικασία αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και όχι μια επίφαση νομοποίησης. Θα είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε όλοι για να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους Ευρωπαίους πολίτες. Ωστόσο, στο βωμό αυτό δεν πρέπει να θυσιάσουμε ένα εξίσου σημαντικό και εκτιμένο των κοινωνιών μας, αυτό της προστασίας των ελευθεριών και των φυσικών προσώπων των προσωπικών δεδομένων. Η ισορροπία είναι λεπτή και τα κοινοβούλια μπορούν να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο εδώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διεύρυνση Περιστατικών Αυθαιρεσία στα σώματα ασφαλεία. Είναι ένα μηχανισμό που θεσπίζεται και ψηφίζεται αυτέ τι μέρε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κλείνοντα, θέλω να αναφερθώ με μία μόνο κουβέντα στου πρόσφυγε, λέγοντα ότι από την Ελλάδα έχουν περάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο προσφύγων και η χώρα μας, η Ελλάδα, παραμένει μια ασφαλής χώρα. Θέλω όμως να τονίσω ότι είναι αναγκαία η στήριξη στο θέμα αυτό των κρατών μελών και όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια και των κρατών μελών να τηρήσουν τι δεσμεύσει του και τι υποχρεώσει του, έτσι ώστε τόσο στα κέντρα υποδοχή, όσο και στα κέντρα που διαμένουν οι πρόσφυγε, να είναι ένα υψηλό επίπεδο φιλοξενία και να μπορούν αυτά να επιτελέσουν το ρόλο τους. Γιατί η κακή εξαθλίωση, η κακή κατάσταση των προσφύγων γεννά εγκληματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And from the European Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τις ομιλήτριές μας, λέει η κυρία Σιλβή Ιβον Κάουφμαν συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Wainwright και συγκεκριμένα. Συζητήσαμε το πακέτο για το άσυλο και εδώ υπάρχει και η νέα εκδοχή του κανονισμού για την Eurodac και έχει ξεκινήσει η κοινοβουλευτική εξέτασή της. Και κατεδείχθη κατά διάφορες συζητήσεις ότι από ό,τι φαίνεται έχει δυσχέρηση η Europol για να έχει πρόσταση στα μητρώα του Eurodac. Ξέρετε ότι γίνεται μέσω εθνικών αρχών. Και συγκεκριμένα είναι η Ολλανδική υπεύθυνη αρχή και τα επίπεδα προστασίας των δεδομένων είναι διαφορετικά. Ερώτημα λοιπόν, μήπως θα μπορούσαμε να το λύσουμε κατά τη γνώμη σας εάν ε, η νέα οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την ε, επεξεργασία ε, για την ε, ε, έρευνα και την προσαγωγή κλιματιών η οποία θα αρχίσει να ισχύει το 2018 και θα μπορούσε ίσως να συνδυαστεί με, τον, με την θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού της Eurodac. Μήπως αυτός ο συνδυασμός θα έλυνε το πρόβλημα λοιπόν για την Europol, για να έχετε πρόσβαση λοιπόν στα μητρώα της Eurodac. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εθνικοί βουλευτές και πάλι. Ο κ. Φερμέλεν από, είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών του Βελγικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Συνάδελφοι, είναι πολύ καλό ότι γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψε με τα εθνικά κοινοβούλια σήμερα γύρω από αυτό το κλασικό θέμα της ε, Europol. Γιατί εξαρτώμεθα ο ένα από τον άλλον, το ένα κράτο μέλο από το άλλο, γιατί η εθνική ασφάλεια του ενό κράτου μέλου συνδέεται άρρηκτα με την εθνική ασφάλεια των υπολείπων. Και η παλιά έννοια του κράτους έθνους του 19ου αιώνα πλέον δεν σταματάει τους ε, τρομοκράτες πουθενά. Επομένω, απαιτείται συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, ε, και γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη μορφή θεραπείας. Και έχετε δίκιο ότι πρέπει να ενισχυθεί η Europol. Υπάρχει νομική πρόβλεψη πλέον να, η Europol να ενημερώνει τους παρόχους για όταν υπάρχουν ε, ε, εγκληματικά εντό αγωγικών tweets και ήδη είπατε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια ε, περιστατικά. Από πού μπορούμε να αντλήσουμε εμεί τέτοια στοιχεία για να ξέρουμε πόσε τέτοιε υποθέσει υπάρχουν και για το κατά πόσο πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή υπάρχει οργανωμένη εκστρατεία από πίσω. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ ε, στην κυβερνοασφάλεια γιατί υπάρχει, υπάρχουν πολλές ε, παράνομες ε, συναλλαγές μέσω του Darknet, του σκοτεινού δικτύου και πώς αυτό συνδέεται με την ε, Θα ήθελα να μας ενημερώσετε. Τέλος, σε ό,τι αφορά ε, τη νομοθεσία για το PNR, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται το Βελγικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή και σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, το Βέλγιο θέλει να ε, επικεντρωθούμε μόνο στα στοιχεία που προκύπτουν και από τις αερομεταφορές αλλά και ε, με τις ε, θαλάσσιες μεταφορές, ε, όλες τις μορφές δηλαδή μεταφορών και θα ήθελα να θέσω τα εξή δύο ερωτήματα. Η Europol πώ ε, θα συμμετάσχει στην ανταλλαγή πληροφοριών PNR και ποια προετοιμασία θα υπάρξει και δεύτερον με ποιον τρόπο μπορεί να εξετάσει η Europol τους τρόπους με τους οποίους ε, οι τρομοκράτες ε, αξιοποιούν τις δυνατότητες μετανάστευσης και τις μεταναστευτικές οδούς για σκοπούς τρομοκρατίας. Κάριον Μίλα από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή Λίμπε και την Τρόικα για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία τη κοινοβουλευτική αυτή συνάντηση, όπου εκπροσωπούνται 23 ε, εθνικά κοινοβούλια, είπατε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 90% των ανταλλαγών πληροφοριών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει από μόνο πέντε χώρε. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη ενισχυμένη συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Είναι λοιπόν αδύρυτη ανάγκη ε, ο Επίτροπος Julian King ε, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν όταν ήταν πρέσβη στη Γαλλία, ε, να στερηθεί και από το κοινοβουλευτικό έργο, το οποίο πρέπει να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό. Για τους σκοπούς της αντιπροσωπευτικότητας του κοινοβουλευτικού, της ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο όλων των συμμετεχόντων είναι κάτι το οποίο μα απασχολεί ιδιαίτερο στη Γαλλία η καταπολέμηση τη δημοκρατίας και την Τετάρτη θα προετοιμάσουμε μια πρόταση, θα παρουσιάσουμε πρόταση ψηφίσματο για αυτό το σκοπό για να διασφαλίσουμε ότι θα συμμετέσχουν και οι γερουσίες ε, ε, των κρατών μελών. Έχουμε λάβει ε, δεν έχουμε λάβει επαρκείς διασφαλίσεις. Έχουμε ακούσει κάποιες δεσμεύσεις, αλλά όχι επαρκείς διασφαλίσεις όπως θα θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε στη νέα οδηγία περί πυροβόλων όπλων. Ε, η Επιτροπή θέλει να απαγορεύσει από οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε χρήση των πυροβόλων όπλων ε, και Υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με τις αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις τρομοκρατικές ενέργειες δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί πυροβόλα όπλα, αλλά όπλα τα οποία αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίου, τα οποία δεν ε, πλήττονται κατά κανένα τρόπο από την ε, νέα αυτή απαγόρευση της Επιτροπής. Προς τον κύριο Wainwright, λοιπόν, θα ήθελα να υποβάλω το εξής ερώτημα. Μπορείτε να μας υποβάλλετε στατιστικά στοιχεία ή αριθμούς σε σχέση με αυτή την ε, εκστρατεία της Κομισιόν κατά των ημιαυτόματων όπλων. Αυτό το θέμα θα απασχολήσει και τα Εθνικά Κοινοβούλια στο Εγγισμέλ. Σινσόφσκι, Βελσέκ, ε, ο οποίος είναι υπεύθυνος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ασφαλείας και μας έρχεται από την Πολωνία. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έγιναν κάποιες γενικόλογες διακηρύξεις, γενικές μάλλον, και φυσικά συμμεριζόμεθα την ικανοποίηση για το ότι του χρόνου θα γίνει άλλο ένα βήμα, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος της Europol. Αυτό θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα ε, τους μεγάλους κινδύνους και τις ε, απειλές που αντιμετωπίζουμε, για παράδειγμα, λόγω της κρίσης του μεταναστευτικού. Σε πολλούς τομείς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προσεκτική στην περαιτέρω ενοποίηση. Αλλά στον τομέα αυτό αξίζει να υπάρξει περισσότερη συνεργασία. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πέρα από τις απειλές στις οποίες αναφερόμεθα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι κίνδυνοι από την σοβαρή εγκληματικότητα για την οποία λέμε λιγότερα. Για παράδειγμα, οι νέες ε, ψυχοενεργές ουσίες, δηλαδή τα υποκατάστατα ναρκωτικών, τα οποία κυκλοφορούν σε πολλά κράτη-μέλη και είναι σοβαρό πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης. Και ξέρω ότι προτείνονται διάφορες ε, λύσεις ε, μέσω ποινικών διαδικασιών στα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν καλό η Europol στα πλαίσια της στενότερης συνεργασίας να ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Ούτω ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόεδρος, η κυρία Κατερίνα Τσίνιτσιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εισηγητές, τους ομιλητές που μας μίλησαν για τις προοπτικές που υπάρχουν για την καταπολέμηση των απειλών κατά των χωρών μας. Πάντα είχα υποστηρίξει την ενίσχυση της Ευρωπόλ, κάτι το οποίο θα αποδώσει καρπούς. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, Επίτροπο τον ε, κύριο Τζούλιαν Κίνγκ γιατί μας μίλησε για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδιαίτερα της τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα ελέγχου ε, δεν θα ελέγχει μόνο την, ε, τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ, αλλά θα ενισχύσει και τη συνεργασία που είναι απόλυτα αναγκαία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και ούτω καθεξής. Έγινε λόγος ήδη σήμερα. Θα ήθελα να σταθώ προσωπικά σε ένα από τα θέματα που έφυξε ο κύριος Wainwright, δηλαδή τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Η Ευρωπόλ είναι εκείνη η οποία έφυξε αυτό το ζήτημα πρωταρχικά. Και ως προς τους ασυνόδευτους λοιπόν ανηλίκους υπάρχει μια δυσκολία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Και φυσικά ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι κατά αυτών των ανηλίκων αφού έχουν ε, διανύσει και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και του κόσμου για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ποιες είναι οι υποδείξεις που θα μπορούσατε να μας κάνετε. Συναδελφοί, έχουμε λίγα λεπτά, αλλά μόνο λίγα λεπτά για να μας απαντήσουν οι ομιλητές. Είναι αδύνατον οι ομιλητές να απαντήσουν σε όλα τα επιμέρους ζητήματα. Ήσασταν όλοι πολύ πειθαρχημένοι, αρκετά πειθαρχημένοι χρονικά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά υπήρξαν και ε, ειδικά ερωτήματα προς τον Ρομπ Βέινραιτ. Και επειδή έχουμε τον ε, επικεφαλής ε, μαζί μας της Ευρωπόλ, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις, απλώς να απαντήσετε σε επιμέρους ε, ζητήματα. Ιδιαίτερα ε, ως προς τα ερωτήματα των εθνικών κοινοβουλίων και ενδεχομένως μπορούν να απαντηθούν και γραπτώς γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, κύριε Κίνγκ, κύριε Επίτροπε, θα θέλατε να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό να έχουμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Πολλά από αυτά τα ζητήματα που καλύψαμε αφορούν δράση των Εθνικών Κοινοβουλίων που βρέθηκαν στο προσκήνιο. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή. Και αυτό είναι και ο απότερος στόχος και ελπίζω να τα καταφέρουμε από κοινού και μέσω της εποπτείας, του μηχανισμού εποπτείας ε, της Ευρωπόλ. Υπάρχουν όμως τομείς όπου η νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Όλοι μας ε, μιλήσαμε για τάχιστη πρόοδο, έτσι ώστε να ε, ολοκληρώσουμε την οδηγία CT και τον ε, κώδικα που αφορά το Σέγγεν και να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των παρανόμων εισαγωγών όπλων. Ελπίζω λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό και τα πυροβόλα όπλα βεβαίως να μπορούν να χρησιμοποιούνται από κυνηγετικού ομίλους, σε αθλητικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Είναι λόγος και για τα προσωπικά δεδομένα και το PNR και πώς μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τον, την άνοιξη του 2018. Επίσης θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση από τα συστήματά μας ως προς την ανταλλογή πληροφοριών. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας πω ότι έχουμε αναλάβει δέσμευση για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος της ιδιωτικότητας. Γιατί πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, αλλά σεβόμενοι απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Επίσης θα πρέπει να επιτελαστεί η εργασία για να καταφέρουμε τα καλύτερα από τις πάρκες πληροφορίες, να ορίσουμε τα κενά, να πληρώσουμε αυτά τα κενά. Θα συναντηθούμε με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων για να συνεχίσουμε τις εργασίες ως προς τις προκλήσεις των συστημάτων πληροφοριών και θα σας ενημερώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, υπάρχει ένα ειδικό ερώτημα ως προς το, τα εγκλήματα στον ε, κυβερνοχώρο. Και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα μέσω εθνικών ε, προγραμμάτων και με βάση εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Επίσης, οφείλω να τονίσω ότι πολύ εκπροσωπείται και το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για την ε, προοπτική, ενδεχόμενη προοπτική αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω το γεγονός ότι η Βρετανική κυβέρνηση επέλεξε και το opt δηλαδή τη συμμετοχή σε αυτό τον κανονισμό, άρα στο εγγύς μέλλον θα συμμετάσχει η κυβέρνηση και σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και στα μέτρα εφαρμογής. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω και όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να προσπαθήσουν να οικοδομήσουμε ε, ένα στεναρό και σταθερό πλαίσιο ασφάλειας και θεωρώ ότι η Ευρωπόλ είναι αναπόσπαστο μέρος. Ο κύριος Μένβρετ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω απευθεία σε ερωτήσει για να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερε. Κύριε Καραμαλή, κ. Και οι δύο αναφέρθηκαν ε, στον ε, μεγάλο αριθμό πληροφοριών ε, που ανταλλάσσονται. Και κάποιο ανέφερε ότι μόλι πέντε κράτη-μέλη είναι αυτά που όντω συμμετέχουν. μπορώ να σα πω με τα χαρά ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση το τελευταίο διάστημα εξαιτία και των αποτρόπων εγκλημάτων σε Βερξέλλε και Παρίσι και πλέον ε, η πλειονότητα των Ελλαδοπών μαχητών που έχουν μεταβεί σε Συρία και Ιράκ έχουν κοινοποιηθεί στι αρχέ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή λοιπόν. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά επίπεδα ανταλλαγής πληροφοριών ε, μεταξύ Europol αλλά και ε, αστυνομικών αρχών και υπηρεσιών ασφαλείας ανά την Ευρώπη. Υπενθυμίζω και αυτό που είπε ο κύριος Μέρα, ότι η Europol πάντα ε, τηρεί τους ε, κανόνες ε, προστασίας δεδομένων με, τρίτες, τρίτα μέρη. Πάντα δηλαδή υπάρχει πρώτερη σύμφωνη γνώμη στην κατάθεση των αρχών για να υπάρξει τέτοια διαβίβαση δεδομένων. Και εγώ συμμερίζομαι τις ε, απόψεις του κυρίου Κίνγκ σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Επέλεξε να κάνει opt-in σε αυτή τη δυνατότητα και εγώ το θεωρώ πολύ καλό. Στο βαθμό λοιπόν που ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, ένα κράτος μέλος πρώτης γραμμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ θετικό αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Διαθεμέρα για τον τρόπο με τον οποίο προώθησε την απόφαση, την πρόταση αυτή έως την τελική της έγκριση. Για την κυρία Γκόμες, όπως ανέφερε για τα έγγραφα Παναμά, η Europol είχε όντως εντοπίσει πολλές διασυνδέσεις ε, δημοσίων πληροφοριών και στοιχείων που υπήρχαν στι δικέ μα ε, βάσει δεδομένων. Έχουμε κοινοποιήσει τι αρχέ. Κανένα κράτο μέλο δεν έχει ζητήσει μέχρι τώρα να ξεκινήσουμε έρευνα. Σε ό,τι αφορά τι ε, νόμιμε και ασφαλεί διόδου, αυτό είναι περισσότερο πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι η θέση μου να απαντήσω η αρμοδιότητα της Europol ή άλλων αρχών επιβολής του νόμου είναι η προστασία των συνόρων μας και να αποτρέψουμε αυτά τα οργανωμένα, μάλλον τα, δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να περνούν τα σύνορα παράνομα και να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Ε, επιβεβαιώνω όντω ότι είναι εξαιρετικό τέρος. η Νορβηγία, τρίτη χώρα. Έχουμε πολυάριθμες συνταλλαγές πληροφοριών κάθε μέρα με πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην πρώτη γραμμή της ε, συνεργασίας αυτής ε, με την ε, Europol. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο που ανέφερε η Ελληνίδα συνάδελφος, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, το κατανοούμε. Σας διαβεβαιώ ότι ο νέος κανονισμός έχει βελτιώσει τα εχέγγυα για την προστασία δεδομένων. Με τον, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων θα έχει σημαντικές και ανεξάρτητες δυνάμεις και εξουσίες για να ελέγχει ακριβώς πώς γίνεται αυτή η συγκέντρωση, συλλογή και αποθήκες για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ε, λογοδοτεί και ενώπιόν σας βέβαια και θα έχει και τη δυνατότητα να δημοσιοποιεί τις ε, εκθέσεις του. Για την κυρία Κάουφμαν και την πρόσβαση ε, στα, στη Eurodac. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο η νέα νομοθετική πράξη 2018 θα είναι η κατάλληλη λύση. Θα πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, όμως και πάλι το θεματολόγιο διαπιστωτικότητας ε, με την Europol θέλει να διασφαλίσει ότι η Europol θα έχει πρόσβαση, αναλογική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για να εξετάσουμε τους τρόπους με τον οποίο οι τρομοκράτε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα δεδομένα. Ο κύριος Βερμέλλον αναφέρθηκε στο Darknet και πώς ε, ε, γίνεται ο πιο εύκολος ε, τρόπος για την ε, διευκόλυνση του οργανωμένου εγκλήματος της τρομοκρατίας στη διαδίκτυο. Εμείς αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα, όμως είναι πολύ δύσκολο να το πράξουμε γιατί για λόγους κρυπτογράφησης είναι πολύ εύκολο για εκείνους να κρύψουν τα ίχνη τους και κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση προσωπικών δεδομένων για να στηρίξουμε κατά το δυνατόν τις αστυνομικές έρευνες. Για το PNR, η Europol έχει αναγνωρισμένο ρόλο στο κανονισμό EUPNR γιατί ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται τα επεξεργασμένα δεδομένα και μεταξύ τους, αλλά και μέσω του μηχανισμού ε, της Europol. Ενθαρρύνουμε λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν ε, το σύστημα της Europol, ούτως ώστε τα επεξεργασμένα δεδομένα αυτομάτως να τη χάνουν ανταλλαγής με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Μιλήσατε και για τις τρομοκρατικές ροές μέσω των μεταναστευτικών ροών. Η Europol για πρώτη φορά έχει φτιάξει δευτεροβάθμια όργανα ε, υποδοχής και εξέτασης θα γίνει αυτό στην Ελλάδα, θα γίνει το ίδιο και στην Ιταλία για να βοηθήσουμε το επιτόπιο προσωπικό ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως για να ταυτοποιήσουμε για να εντοπίσουμε τυχόν προσπάθειες τρομοκρατών να εισέλθουν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τέλος, κύριο Χαλαιοάνο και πιο συγκεκριμένα για τα πυροβόλα όπλα. Εδώ δεν έχουμε ε, στοιχεία που να καταδεικνύουν την χρήση τέτοιων νόμιμων πυροβολών όπλων από τρομοκράτε. Όμω μπορώ να πω ότι η στρατηγική που προτείνεται μέσω και τη προτείνομενης οδηγία είναι να μην αφήνουμε πλέον περιθώριο Στου τρομοκράτε και εγκληματίε, να έχουν πρόσβαση σε τέτοια πυροβόλα όπλα με οποιοδήποτε τρόπο. Και ξέρουμε ότι τέτοια ε, κλεμμένη πυροβόλα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε τετοιε επιθέσεις. Δεν είναι βέβαια, ε, δεν φταίνε οι ιδιοκτητε των ε, όπλων αυτών, ομω είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Υπενθυμίζω και αυτό που ανέφερε ο Επίτροπος, ότι η οδηγία έχει ως σκοπό, αφορά μάλλον ε, τα αυτόματα ή αυτόματα όπλα στρατητικού τύπου. Και θέλουμε αυτό να περιοριστεί μόνο στις ε, αθλητικές καταστάσεις και, και τα λοιπά. Θέλουμε λοιπόν να μην αφήνουμε πλέον περιθώριο στους ε, τρομοκράτες και εγκληματίες να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα πυροβόλων όπλων γιατί βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει και εξελίξει στους τρόπου που χρησιμοποιούν πλέον οι τρομοκράτε. Αν έχω ξεχάσει κάτι, μπορούμε να τα απαντήσουμε και μέσα από τι διαδικασίε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ανέφερα αυτή τη δυνατότητα, συνάδελφοι, ο πρόεδρο, γιατί σε πολλέ τέτοιε διακοινοβουλευτικέ συναντήσει, όπω ξέρουν και οι συνάδελφοί μου, πολλοί δεν ικανοποιούνται από τι απαντήσει. Γιατί υπάρχουν εδώ συνάδελφοι από επιτροπέ ε, εσωτερικών, από επιτροπέ ε, νομικών θεμάτων. Υπάρχουν πολλέ ερωτήσει που θέλετε να θέσετε στον Επίτροπο και τον κεφαλή τη Europol. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλέ άλλε αναλυτικέ ερωτήσει που θα μπορούσατε να θέσετε. Αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει χρόνο. Αν υπάρχουν λοιπόν. Εντάξει, τώρα έχετε έρθει σε επαφή με τον άλλον. Αν υπάρχουν άλλε ερωτήσει, παρακαλώ, ε, στείλτε σε εμά, στη γραμματεία μα, να τι στείλουμε στη Europol και στον κύριο Επίτροπο, γιατί νομίζω ότι και από ε, συμβολική αλλά και από ουσιαστική πλευρά έχει μεγάλη σημασία να έχουμε αυτές τις απαντήσεις αυτές τις πολύ συγκεκριμένε όπως είδαμε ερωτήσεις. Τέλος, να δώσω το λόγο <clears throat> για δύο τελικά λόγια παρακαλώ αν θέλετε στον κύριο Αμπό παρακαλώ Ευχαριστώ Πρόεδρε Ρωτήθηκα αν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το PNR θα λειτουργήσει απόλυτα αποτελεσματικά. Προφανώς κανένα σύστημα δεν ε, εγγυάται αποτελεσματικότητα 100%. Προσπαθούμε τώρα να στήσουμε ένα σύστημα. Και νομίζω ότι αναφέρθηκαν και οι δύο πλευρέ. Από ότι μία πρέπει να είναι αποτελεσματικό το σύστημα, πρέπει να υπάρχει διεθνή συνεργασία, αλλά παράλληλα και είναι εξίσου σημαντικό πρέπει να σεβαστούμε τις δημοκρατικές μας παραδόσεις. Έλεγχος επί μια αστυνομική δραστηριότητας, ούτω ώστε να εγγυώνται οι δημόσιες ελευθερίε. Αυτή η ισορροπία, αυτή η ε, πράξη ισορροπισμού, αυτή είναι σημαντική. Ευχαριστώ, ο Έληξε αυτή η πρώτη συζήτηση. Καταληκτικά θέλω να πω, όπως ε, δεν είπα επαρκώς στην αρχή, ότι το γεγονός ότι μπαίνουμε σε νέα φάση της ε, Ένωσης Ασφάλειας σημαίνει ότι εμείς ως ευρωβουλευτές προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις κύριες γραμμές αυτής της Ένωσης Ασφάλειας. Όπως μας είπε και ο Επίτροπος, θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερος ρόλος για τους ε, ειδικού φορείς, αλλά κάτι άλλο πρέπει να αναφέρω, ότι ως Κοινοβούλιο ασχολούμεθα με την οδηγία κατά της τρομοκρατίας, μόλις την ολοκληρώσαμε, έχουμε ένα ε, μπουκέτο νομοθετημάτων που εντάσσονται στον τομέα αυτό. Αλλά θέλουμε να υπάρξει και εφαρμογή αυτών που αποφασίζουμε. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Κίνγκ θεωρεί ότι είναι βασική προτεραιότητα. Δεν έχει καμία έννοια να υπάρχει νομοθεσία για την ασφάλεια αν δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να σας δώσουμε ως Ευρωβουλευτές. Όταν ε, ε, για παράδειγμα συζητάμε για την ε, λεύκανση προϊόντος εγκλήματος, για PNR, αντιτροποκρατία, θέλουμε να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Όταν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, μετά πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δική τους. Και ξέρω ότι αυτό σας απασχολεί σας ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν ερώτημα για όλους μας αυτό. Και μερικοί συνάδελφοι είναι υπεύθυνοι για τέτοια θέματα. Όπως ε, είπε και ο κύριος Δίαθ Δεμέρα, ο κανονισμό της Europol. Και αυτός πρέπει να εφαρμοστεί. Ήθελα να το αναφέρω. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους ομιλητές μας, τον Επίτροπο King, τον Sir Julian King, τον Βουέιν Wainwright, ε, επικεφαλής της Europol και τον Ντομιγίν Ραμπέργκ της Επιτροπής ε, ε, Συνταγματικών Θεμάτων, Νομοθεσίας και Διοικητικών Θεμάτων της Γαλλικής Εθνικέλευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στη δεύτερη συζήτηση και παρακαλώ τους ομιλητές για τη δεύτερη να ανέβουν στο βήμα εδώ στο Προεδρείο και όσο ανεβαίνετε για να μην χάσουμε χρόνο να παρουσιάσω το θέμα μας όσο αλλάζουν εδώ οι συγκαθήμενοι μου. με συγχωρείτε που δεν υπάρχει διάλειμμα. Θα συνεχίσω. Και σας παρακαλώ ελάτε εδώ στο Προεδρείο όσο πιο σύντομα γίνεται. much time for selfies and, uh, Παρακαλώ δεν υπάρχει χρόνος για selfie και διάφορα άλλα. Λοιπόν, εντάξει, okay. Ε, ε, θα κάνω μια σύντομη διακοπή για να έρθουν εδώ οι μιλητές. Um, λοιπόν, συνάδελφοι, λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται το χρόνο μας. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Λοιπόν, συνάδελφοι, λοιπόν, τώρα θα διεισδύσουμε σε βάθος στο θέμα του ελέγχου της Europol. Το κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, του φορέα αυτού. Η δεύτερη συνεδρίασή μας ασχολείται με τις πρακτικές λεπτομέρειες για την ομάδα κοινού κοινού κοινοβουλευτικού ελέγχου που ε, εγκαθιδρύεται με βάση τον νέο κανονισμό του Europol. Όπως ξέρετε, η διάσκεψη Προέδρων των ε, Κοινοβουλίων της Ένωσης συμφώνησε τον περασμένο Μάιο μια σταδιακή προσέγγιση για να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργία αυτής της κοινή κοινοβουλευτικής ε, ομάδας ελέγχου συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης μια διακοινοβουλευτικής συνάντησης για να μας εξηγηθεί περαιτέρω αυτή η σταδιακή προσέγγιση και τι έχει γίνει μέχρι τώρα Χαίρομαι που θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Εντίτα Φάντναρ, που είναι η συγγήτρια τη Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου τη Σλοβακική Δημοκρατία για Ευρωπαϊκέ Υποθέσει για θέματα δικαιοσύνη και εσωτερικών. Επίση, είναι επικεφαλή τη ομάδα εργασία τη Τρόικα για τι λεπτομέρειε του Europol. Δηλαδή, τι πρακτικέ λεπτομέρειε λειτουργία. Modalities στα αγγλικά. Η Τρόικα τώρα αποτελείται από το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία, την Εστονία και συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Φούντνερ, εμεί θα μα εξηγήσετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και την προσέγγιση σα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συναδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που οργάνωσε αυτήν την διακοινωνιστική συνάντηση για την Europol και που δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός για την ε, κοινή διαδικασία ελέγχου της Europol. Να σας ενημερώσω γιατί τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Τρόικα. Όπως ξέρετε, η ομάδα εργασίας της Τρόικα αποτελείται από εκπροσώπους της Εστονίας, του Λουξεμβούργου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Δημιουργήθηκε με εντολή να καθορίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες της ομάδας κοινού, κοινού κοινοβουλευτικού ελέγχου με βάση τα απορίσματα της συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων του Μαΐου 16 στο Λουξεμβούργο. Οι πρόεδροι των Κοινοβουλίων συμφώνησαν σε μια σταδιακή προσέγγιση. Το πρώτο βήμα ήταν να υπάρξει μια διαβούλευση όλων των νομοθετικών σωμάτων της Ένωσης. Ευθύς εξ αρχής η ομάδα εργασία συμφώνησε ότι οι λεπτομέρειες αυτής της ομάδας κοινού ελέγχου πρέπει να καθοριστούν πριν ε, αρχίσει να ισχύει ο νέος κανονισμός της Europol, δηλαδή πριν την 1η Μαΐου. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε αποφασίσει την ε, σύνθεση τον τρόπο λειτουργίας και προεδρίας και τον ε, τόπο λειτουργίας αυτού του σώματος αυτού. Στείλαμε λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα νομοθετικά σώματα της Ένωσης την 1η Σεπτεμβρίου. Περιείχε κυρίως τρία ερωτήματα για τις τρεις κύριες πρακτικές λεπτομέρειες και ένα επιπλέον θέμα που είχε να κάνει με την εμπειρία των ε, νομοθετικών σωμάτων για τον έλεγχο αρχών επιβολής του νόμου. Ανταποκρίθηκαν 34 νομοθετικά σώματα από 25 κράτη-μέλη της Ένωσης <clears throat> και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομάδα εργασίας εξέτασε αναλυτικά όλες τις ε, αντιδράσεις όπως ξέρετε με βάση την τεκμηρίωση που έχετε στη διάθεσή σας, οι αρχικές απαντήσεις ήταν ε, πολύ διαφορετικού χαρακτήρα αντανακλώντας μια ευρία γκάμα απόψεων των ευρωπαϊκών νομοθετικών σωμάτων για τους βασικούς κανόνες λειτουργίας αυτής της ομάδας. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις για τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Προσπαθώντας να βρούμε μία μέση οδό. Και ασχοληθήκαμε και με γενικότερε παρατηρήσεις των κοινοβουλίων για την αποτελεσματικότητα, την ισορροπία, την ισονομία και τα κύρια καθήκοντα. Οι συμβιβασμοί μα βασίζονται στι ε, ε, σχετικές διατάξεις του νέου κανονισμού τη Europol. Οι διατυπώσει των συμβαστικών προτάσεων σα απεστάλησαν στι 25 Νοεμβρίου και θα είναι το κύριο κείμενο για τι σημερινέ μα συζητήσει να σας παρουσιάσω τις ε, μεμονωμένες συμβαστικές προτάσεις για την συμμετοχή σε αυτή την ομάδα. Τα αγγλικά αρχικά είναι JPSG. Οι αντιδράσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και άλλων σωμάτων δεν έχουν δείξει σαφή προτίμηση για καμία εναλλακτική λύση. Ορισμένα νομοθετικά σώματα θεωρούν ότι διάφορες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Οπότε εμείς ως συμβασμό προτείνουμε τα μέλη αυτά να ορίζονται ατομικά από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η σύσταση είναι τα μέλη να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία και να συμμετέχουν στις ε, σχετικές επιτροπές ή υποεπιτροπές των Εθνικών Νομοθετικών Σωμάτων. Έτσι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι διαφορέ προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών σωμάτων και θα έχουμε δυνατότητα να ωφεληθούμε από τι γνώσει. Για τον αριθμό. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν μα έδωσαν σαφή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ε, προτείνουμε διάφορες μορφές διακοινοβουλευτική συνεργασία. αλλά τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια δεν επέλεξαν καμία από τις υπάρχουσες μορφές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και προτίμησαν μια νέα δομή. Καταλήγουμε λοιπόν ότι θα είναι αναγκαίο να βρούμε μια εντελώς νέα δομή για αυτό το JPSG. Ορισμένα εθνικά νομοθετικά σώματα θεωρούν ότι η αριθμητική σύνθεση αυτής της ε, ομάδας πρέπει να καθοριστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά το JPSG και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, συστήματα δύο νομοθετικών σωμάτων. Συγκεκριμένοι αριθμοί τώρα. Διαπιστώσαμε ε, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων προτάσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται από ένα έως έξι μέλη το καθένα. Γιατί προτείνουν ε, ε, και διαφορετικές ε, προσεγγίσεις για την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλοι προτείνουν μονομένα μέλη και άλλοι λένε ότι πρέπει να συμμετάσχει ολόκληρη η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συζητήσαμε ως ομάδα την, ε, τον αριθμό μελών προσπαθώντας να επιτύχουμε ένα συμβασμό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα να λειτουργεί αποτελεσματικά και να εξισορροπεί την εκπροσώπηση των ε, Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και τον νέο κανονισμό της Europol. Λόγω της περιπλοκότητας του θέματος αυτού, χαίρομαι που η ομάδα εργασίας κατάφερε να καταλήξει σε ένα λογικό συμβιβασμό. Η πρότασή μας είναι να, να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε χώρα. Εάν έχουμε δύο νομοθετικά σώματα σε κάποιο κράτος, θα είναι ένα από κάθε νομοθετικό σώμα και 6 εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε ο συνολικό αριθμό θα ήταν 62. Η ομάδα εργασία μα θεωρεί ότι αυτή η πρόταση επιτυγχάνει την ε, σωστή ισορροπία εκπροσώπησης μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν ευνοείται ούτε η μία, η πλευρά των Εθνικών, ούτε η άλλη, η πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο αριθμός είναι σχετικά μικρός, 62. Και νομίζουμε ότι είναι σωστός αριθμός για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία και να αντιμετωπίζει τα πολύ ουσιώδη θέματα που θα έχει ενώπιόν της αυτή η ομάδα. Όσον αφορά την Προεδρία, τον τόπο και την ε, περιοδικότητα συναντήσεων, λάβαμε πολλές απαντήσεις. Πολλά εθνικά κοινοβούλια θεωρούσαν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει λειτουργικότητα αλλά και η σωστή αξιοποίηση των πόρων. Αναλύοντας τις απαντήσεις ε, υποδιαιρέσαμε το θέμα σε μια σειρά από υποθέματα. Τα περισσότερα κοινοβούλια θεωρούν ότι η προεδρία της ομάδας αυτής πρέπει να αναλαμβάνεται από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δημοβουλίου και εκπρόσωπο τη εναλλασσόμενη Προεδρία τη Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι συμβατό με τον κανονισμό τη Europol επίση. Ε, τέθηκε το θέμα πόσο τακτά πρέπει να συνεδριάζει αυτή η ομάδα, η ομάδα εργασίας μας, εξέτασε και τον κανονισμό και προτείνει ότι Βλέποντας ότι είναι περιορισμένη χρονικά η λειτουργία της ομάδας μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεδριάζει για να συζητάει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Europol. Τα άλλα καθήκοντα συνάντηση με τον επικεφαλής της Europol δεν είναι περιορισμένα όμως χρονικά. Λόγω αυτού και επειδή ορισμένα εθνικά κοινοβούλια θεωρούν ότι πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά αυτή η ομάδα, προτείνουμε η ομάδα να συναντάται μια φορά το χρόνο και αν είναι αναγκαίο να μπορεί σε αυτή τη συνάντηση να συζητά για αρκετές μέρες. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συμπρόεδρος θα μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτες συνεδριάσεις. Για να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα η ομάδα μας η ομάδα εργασία πρότεινε η ετήσια τακτική συνεδρίαση της ομάδας αυτής, του JPSG, να γίνεται στις Βρυξέλλες και έκτακτες συναντήσεις να μπορούν να λάβουν χώρα στη χώρα της Προεδρίας της Ένωσης. Ε, με τη συνένεση βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνάδελφοι μου και εγώ περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας επί των ε, προτάσεων μας αυτών Σύμφωνα με τα πορίσματα των Προέδρων των Κοινοβουλίων, οι προτάσει σα θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη πρότασή μα, την οποία θα στείλουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου τρέχοντος. Τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017. Κατόπιν, η τελική διατύπωση θα εγκριθεί στην Μπρατισλάβα στις 23 και 24 Απριλίου στη διάσκεψη των Προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτά προς το παρόν και προσλέπω στην περαιτέρω συζήτηση επειδή πρέπει να επιστρέψω για κάτι ιδιαίτερα επίγον στην ε, Σλοβακία θα χρειαστεί να αποχωρήσω στις 5 περίπου αλλά οι συνάδελφοί μου θα σας ακούσουν πολύ προσεκτικά και θα με ενημερώσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε όλο το σχέδιο πρότασης, έχει διανεμηθεί και θέλουμε να ακούσουμε τις αντιδράσεις σας. Καταρχήν θα ακούσουμε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κύριο Ντίας Ντεμέρα, ο οποίος ήταν βασικός συγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ε, κανονισμό της Ευρωπόλ. Κύριε Ντίας Ντεμέρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους ε, συναδέλφους του δεύτερου αυτού πάνελ. Θα δώσω ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με αυτά που προείπε η Σλοβακική Προεδρία, που νομίζω ότι είναι χρήσιμες για να ενισχύσουμε τη συζήτηση στη συνέχεια. Τώρα, ως προς ε, ορισμένα νεότερα, γενικού περιεχομένου, η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου υποβλήθηκε με ένα πρώτο το κείμενο ενός, ε, της, της Μικτής Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τον Ιούνιο του 2013. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι για 7 χρόνια εργαστήκαμε στα πλαίσια της ε, Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Ε, εγώ ήμουν εισηγητής με βάση την απόφαση του Συμβουλίου και έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που ισχύει τώρα. Τώρα θα αντικατασταθεί από έναν κανονισμό που θα ισχύει από την 1η Μαΐου του 2017 και θα διέπει όλες τις ε, λειτουργίες και αρμοδιότητες της Ευρωπόλ. Λάβαμε υπόψη τις υποδείξεις που έγιναν και από πλευράς ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε συζητήσεις με τη Βουλή των Λόρδων και έγινε λόγος και για το άρθρο 51 του κανονισμού της Ευρωπόλ, με βάση το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα ορίσουν από κοινού την οργάνωση και σε μερικούς μήνες θα συντάξουμε και τον ιστορικό κανονισμό της ε, μικτής ομάδας δυνάμει του άρθρου 9 του πρωτοκόλου υπαριθμών 1. Όπως ε, προείπα, στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους ε, εγκρίθηκε το πλαίσιο και θα ισχύσει από τον Μάιο του 2017. Ορίζεται λοιπόν ένα πλαίσιο λειτουργίας για τα πιο βασικά ζητήματα της ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου και υπάρχουν ορισμένα σημεία κλειδιά στα οποία αναφέρθηκε η Σλοβακική Προεδρία όπως η σύσταση, η Προεδρία και η έδρα καθώς και ο τόπος συνεδριάσεων. Μιλήσαμε για τη συμμετοχή τριών κοινοβούλιων, μάλλον τρία κοινοβούλια, εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Και στη συνέχεια θα φτάσουμε σε μια συμφωνία, σε ένα προσχέδιο συμφωνίας για να είμαι πιο ακριβής σε σχέση ε, με την επόμενη διάσκεψη των εκπροσώπων στη Βρατισλάβα στις 24-25 ε, Απριλίου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη αυτό το χρονοδιάγραμμα γιατί θα πρέπει να συνέλθουμε με βάση το πλαίσιο που μας διέπει μέχρι την 1η Μαΐου. Μιλήσαμε λοιπόν για το σημαντικό ρόλο της Ευρωπόλ και λαμβάνοντας υπόψη και τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπόλ, δηλαδή την τρομοκρατία, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, δραστηριότητα της Ευρωπόλ, την αστυνομική εποπτεία σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη. Εγώ ως εισηγητής της απόφασης και τώρα του κανονισμού πάντα έδειξα μεγάλη εμπιστοσύνη στην εργασία του οργανισμού και είχα και την δυνατότητα να ελέγξω τις δραστηριότητες του στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι και εγώ συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ μεταξύ 2002 και 2004, εκπροσωπώντας το βασίλειο της Ισπανίας. Φυσικά η Ευρωπόλ ε, δεν ε, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να προασπίσει την χρήση των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό χρειάζεται ένα εύρωστο σύστημα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το άρθρο 88 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει το εξής. Η διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ θα διεκπεραιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό η πρόταση της Επιτροπής του 2013 ε, δεν ήταν ε, πλήρης και γι' αυτό ε, προώθησα την τροπολογία υπαριθμών 200 όπου γίνεται λόγος για την εφαρμογή του άρθρου 88 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος από εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα εθνικά. Και η Ευρωπόλ πρέπει να ενισχύσει τα κράτη-μέλη στη δραστηριότητά τους, διότι η δράση της βασίζεται στις υποδείξεις των κρατών μελών, γι' αυτό είναι αναγκαίος ο κοινοβουλευτικός αυτός έλεγχος. Ο νέος αυτός έλεγχος λοιπόν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δηλαδή την εμπιστοσύνη για, να, για την αποκοινού συμμετοχή. Αυτό ήταν ένα από τα δύνατα σημεία της Ευρωπόλ στο παρελθόν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο συνεργατικοί στον τομέα της πρόληψης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά κατά τις διαπραγματεύσεις για να πείσουμε το Συμβούλιο και να θέσουμε σε εφαρμογή έναν επαρκή και λειτουργικό μηχανισμό ελέγχου. Τώρα, σε σχέση με τον προσδιορισμό των μελών, την σύνθεση, την προεδρία ε, τον τόπο συνεδρίασης και τον αριθμό των συνεδριάσεων, θα πρέπει να πω τα εξής. Για εμένα ως εισηγητή, Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή η μεικτή ομάδα να είναι μικρή, ευέλικτη, εξειδικευμένη και αποδοτική. Να έχει ένα ελεγχόμενο μέγεθος. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι το άρθρο 88 δεν ορίζει αναλογικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών. Το μόνο που ορίζει είναι ίση συμμετοχή, ισότητα στη συμμετοχή. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εμπειρογνώμονες επί του θέματος είδαμε στα, στις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια θέσεις που αναφέρουν ότι σε αυτό τον ε, ε, μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου θα μπορούσαν να συμμετέχουν και ε, φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ε, εμπειρογνωμοσύνης, πραγματογνωμοσύνης. Και βεβαίως θα υπάρχει και ένα θέμα εκπεριτροπής ε, ανάληψης καθηκόντων. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει για να είμαστε αποδοτικοί να υπάρχει μια σταθερή γραμματεία και φυσικά η έδρα να είναι αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για οικονομικούς και επιμελητιακούς λόγους και για λόγους ε, ε, παροχής υπηρεσιών διερμηνίας και ούτω καθεξής. Θα μπορέσουμε να έχουμε έναν δημοκρατικό και πραγματικό έλεγχο της Ευρωπόλ, ο οποίος δεν θα είναι ελλειπής γιατί φτάσαμε σε έναν ρεαλιστικό συμβιβασμό μεταξύ ημών. Εγώ είμαι αλληλέγγυος με την Τρόικα σε σχέση με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου σε, αυτής, σε αυτές τις συστάσεις. Βεβαίως, έχω τις επιφυλάξεις μου και θα τις εκφράσω κατά τη διάρκεια των μελλοντικών συζητήσεων. Σήμερα μου ελέγχθη ότι ένα κράτος μέλος θα υποβάλει τροπολογίες. Μα αυτή είναι και η διαδικασία που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Και εγώ θα υποβάλω τροποποίησης και προτάσεις τροπολογίας. Σε σχέση τώρα με τα καθήκοντα, όπως είπε και η Σλοβακική Προεδρία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων έχουν οριστεί από το άρθρο 51 της Συνθήκης της Ευρωπόλ. Θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα αυτό το σημείο, ότι θα ήθελα ε, να ε, αδράξω την ευκαιρία της ε, παρουσίας σας να μιλήσω και για τη συμμετοχή του Ισπανικού Κοινοβουλίου που ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Δίας Σταμέρα. Συνάδελφε, θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα. Όχι. Συνέχεια. Στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανάλυση και για την επικοδομητική κριτική σας επί της πρότασης ήταν ε, πολύ χρήσιμη. Στο γεμικό σχήματος θα ακούσουμε τώρα την κυρία Νίτα Σάφερ να μας δώσει την ε, οπτική γωνία της Bundestag από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα συναντηθήκαμε για να θέσουμε τη βάση ενός νέου οργάνου ελέγχου της Europol από τα κοινοβούλια μας. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντική η λειτουργία αυτής της αρχής, σε αυτή τη συγκυρία. Και γι' αυτό αυτή η νέα φάση διακοινοβουλευτικής συνεργασίας θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρή. Θεωρώ ότι είναι κοινό μας καθήκον να εφαρμοστεί και να διαμορφωθεί όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ούτως ώστε να επιτύχει, να συμβάλλουμε στην επιτυχία της Europol. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια από κοινού θα κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο μιας ε, Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Αρχής. Είναι ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, ιστορική σημασία βήμα κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Μέχρι στιγμής η διακοινοβουλευτική μας συνεργασία είναι κυρίως ε, κάποιες συνεδριάσεις, ε, για παράδειγμα με βάση το άρθρο 13, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Οπότε από πλευρά των συναδέλφων μου από το γερμανικό Bundestag θέλω να ευχαριστήσω την Τρόικα και ιδιαίτερα την Σλοβακική Προεδρία για την εξαίρετη προπαρασκευαστική εργασία με τις διαβουλεύσεις που κάνανε των κοινοβουλίων και με τις προτάσεις που υπέβαλαν βοήθησαν την ανταλλαγή απόψεων και την κατανόηση και συμφωνία για την, ε, το μέλλον αυτού του οργάνου. Ευχαριστώ επίσης για την ευκαιρία που υπάρχει για να υποβάλει η Γερμανική Βουλή περαιτέρω προτάσεις για τη λειτουργία αυτού του οργάνου και για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση. Ευχαριστώ επίσης όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, τα οποία υπέβαλαν ε, πολλές καλές προτάσεις μέσω της ανταλλαγής αυτών, αυτής των ερωτηματολογίων και μέσω της πολυπληθούς συμμετοχή του σήμερα. Από πλευράς Bundestag ευχαριστούμε πολύ την Τρόικα και την πρόταση που κάνει, ούτω ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να επιλέξουν τους εκπροσώπους αυτήν την ομάδα από τους πιο ειδήμονες και από τις ειδικέ επιτροπές. Προτείνουμε επίσης τα μέλη αυτής της αρχής να εκλέγονται για τη διάρκεια της εντολής των Εθνικών Κοινοβουλίων, ούτω ώστε να μπορέσουν να δώσουν τη γνώση τους και να υπάρχει μια συνέχεια, να υπάρχει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Τα μέλη αυτής της ελεγκτικής αρχής πρέπει να γνωρίζονται μεταξύ τους και να μπορούν από κοινού να ανταλλάσσουν και να συλλέγουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους. Όσον αφορά την τακτικότητα των συνεδριάσεων, η Τρόικα προτείνει μία συνεδρίαση το χρόνο. Και αν υπάρχει ανάγκη, θα μπορούσε να ε, λάβει η χώρα μια δεύτερη συνεδρίαση. Πάνω από τα μισά εθνικά κοινοβούλια, μεταξύ των οποίων και το γερμανικό, εκφράστηκαν για ε, δύο φορές το χρόνο συνεδριάσεις. Αυτή η περιοδικότητα έχει να κάνει με το χαρακτήρα των καθηκόντων και με την ανάγκη ε, ελέγχου μετά την ε, θέση σε ισχύ του κανονισμού. Οι υπάρχουσες συναντήσεις μέχρι τώρα, όπως η ΚΟΖΑΚ και ε, άλλες τέτοιες όπως το 2013, πρέπει να είναι το παράδειγμα. Πρέπει και εμείς όπως και εκείνοι να μπορούμε να συνεδριάσουμε και αν υπάρχει ανάγκη θα πρέπει να, να μπορούν να γίνουν και έκτακτες συνεδριάσεις. Για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία του οργάνου θα είχε έννοια να υπάρχουν και ομάδες εργασία για επιμέρους ειδικά θέματα, εάν χρειαστεί. Όλοι μας ε, οι κόποι είναι για να υπάρξει αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου αυτού, για να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία της Europol. Γι' αυτό ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι σημαντικό θέμα. Η Τρόικα προτείνει δύο αναεθνικό κοινοβούλιο ή ένα ανανομοθετικό σώμα, υπάρχουν δύο νομοθετικά σώματα, συν έξι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως για να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη την σύνθεση των Ευρωπαϊκό, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εθνικού Κοινοβουλίου οποιαδήποτε απόφαση. Μέσω των απαντήσεων καταδεικνύεται μια πλειοψηφία για να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις εκπρόσωποι ένα Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτή η θέση περιέχεται και στη θέση της Γερμανικής Βουλής. Πρέπει να κάνουμε μια πρώτη σε βάθος συζήτηση για τα θέματα αυτά και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από τον αριθμό των μελών, αλλά από τους στόχους που θα τεθούν και από τον τρόπο εργασίας του σώματος αυτού. Και αυτά τα θέματα πρέπει να τα συζητήσουμε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ τώρα σε κάποια περαιτέρω θέματα, τα οποία δεν ήταν εκπεφρασμένος ε, περιεχόμενα στο ερωτηματολόγιο, αλλά που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δράσουμε σύντομα, γιατί ο νέος κανονισμός της Europol θα αρχίσει να ισχύει την 1η Μαΐου 17. Γι' αυτό προτείνω να συζητήσουμε και περαιτέρω θέματα μέχρι τότε του τρόπου λειτουργίας. Μόνο έτσι μπορούμε τάχιστα μετά την σύσταση να αναλάβει τα καθήκοντά της αυτή η ομάδα και να επιτελέσει το έργο της. Να μην κάνουμε το σφάλμα όπως έχει γίνει για άλλες ε, μόνιμες ε, διακοινωνιστικές δομές, να συζητάμε για δύο χρόνια για οργανωτικά θέματα από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σώμα, γιατί δεν θα έχουν επιληθεί εκ των προτέρων. Γι' αυτό το λόγο η Γερμανική Βουλή προτείνει να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση. Και θέλω να την ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Το θέμα της ε, σύστασης του σώματος για να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία πρέπει να διευκρινιστεί. Και πρέπει να διευκρινιστεί και ο τρόπος ε, ψηφοφορίας και η απαρτία. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά τα θέματα θα μπορέσουν να αποφασίζονται μόνο στις τακτικές συναντήσεις και μάλιστα με τρόπο συναντικό. Επίσης, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να καταστούν σαφώς οι αρμοδιότητε αυτή τη αρχή μεταξύ των συνεδριάσεων του. Δηλαδή, θα μπορούσαν τα μέλη να στέλνουν ερωτήματα στο Διευθυντικό Συμβούλιο τη Europol. Επιπλέον, Πώ θα συνεργαζόμεθα με άλλα ευρωπαϊκά σώματα. Για παράδειγμα, τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Frontex, και πρέπει να επιληθούν και οργανωτικά θέματα. Για παράδειγμα, θα υπάρξει μια γραμματεία και πώς θα αποτιμώνται οι πληροφορίες και εκθέσεις που θα λαμβάνει το σώμα αυτό με βάση το κανονισμό της Europol και η προετοιμασία των πορισμάτων της εργασίας. Αυτό σημαίνει μόνιμη εργασία αυτής της Επιτροπής και μόνιμη κοινοβουλευτική διεύθυνσή της. Αλλά χρειάζεται και διοικητική υποστήριξη. Με βάση την πείρα δημιουργία άλλων διακοινοβουλευτικών σωμάτων πρέπει να σκεφτούμε πώς θα καθοδηγήσουμε ταχαίως την διαδικασία ενώπιών μας. Και αναφέρομαι στην σύσταση της Τρόικα η συνεδρίαση η σύσταση σε σώμα του σώματος να γίνει τάχιστα ούτω ώστε να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί το δεύτερο εξάμεινο του 17 αυτό το σώμα. Άρα από εμά πλέον εξαρτάται να θέσουμε και να στείλουμε τα σωστά μηνύματα για τη λειτουργία του σώματος να επιτύχουμε συνένεση με βάση τις προτάσεις της Τρόικα και να αντιμετωπίσουμε τα περαιτέρω επίγοντα θέματα. Ήδη τώρα. Γιατί οι προτάσεις της Τρόικα τα μέσα Δεκεμβρίου πρέπει να αποτελέσουν μια στέρη βάση για να δημιουργηθεί και να έχει τρόπο λειτουργίας αυτή η νέα διακοινοβουλευτική δομή, ούτως ώστε η διάσκεψη των Προέδρων το 2017 να επιτύχει ένα στόχο και για να μπορέσει το σώμα αυτό να αρχίσει να λειτουργεί. Επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρομοκρατία και οργανωμένη εγκληματικότητα, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δράσουμε. Και νομίζω ότι και κατά την πρώτη συζήτηση ε, τονίστηκε σαφώς αυτό από πλευρά του Bundestag. Σας δηλώνω ότι είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να συνεργαστούμε ενεργά για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σάφερ. Δύο ομιλητές μας μένουν ακόμα πριν ε, ανοίξει η συζήτηση στα υπόλοιπα μέλη. Hans Born είναι ο επόμενος ομιλητής, ερευνητικό τμήμα του Ελβετικού Κέντρου Δημοκρατικού Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει ε, κάνει πολλές δημοσιεύσεις σε ό,τι αφορά τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κοινοβουλευτικού ελέγχου σε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 είναι διεθνής οργανισμός βάσει του ελβετικού ε, δικαίου και έχουμε 65 ε, κράτη που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε συνεργαστεί ανατακτά χρονικά διαστήματα και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενισχύσουμε τις δυνατότητες όλων των φορέων και σε εθνικό επίπεδο και για να εικονίσουμε έρευνα για το πώς ε, μπορούν αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί να επιβλέπουν ε, τις εθνικές αστυνομικές αρχές. Η κοινή κοινοβουλευτική ομάδα, συγγνώμη, ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως προτείνεται από την Τρόικα, συμπεριλαμβάνει 62 μέλη, 56 από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξι από τον ΕΟΚ. Βεβαίως θα υπάρχει η πολυμορφία μεταξύ κρατών μελών. Οι τρομοκρατικές απειλές ε, για τις χώρες της Βαλτικής διαφέρουν πολύ από τις απειλές ε, για την ασφάλεια της ε, Πορτογαλίας και αυτές με τη σειρά διαφέρουν από τις τρομοκρατικές απειλές στην Ελλάδα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την πρόσβαση στι ε, διαβαθμισμένε πληροφορίε. Όπω και εδώ στο Κοινοβούλιο δεν έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση σε ευαίσθητε πληροφορίε. Γι' αυτό η πολυμορφία θα υπάρχει θα το αποδεχθούν αυτό και τα μέλη και νομίζω ότι το σημείο εστίαση θα είναι κυρίω τα στρατηγικά και όχι τα επιχειρησιακά ζητήματα. Στρατηγικά ζητήματα, για παράδειγμα, ποιε πρέπει να είναι οι προτεραιότητε τη Europol. Τι μορφή θα πρέπει να λάβει η οργάνωσή τη, τι προπολογισμό θα λάβει, σε τέτοιο επίπεδο δηλαδή. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό αυτή η ομάδα ε, να συσταθεί. Και συμφωνώ με την κυρία Σέφερ ότι για πρώτη φορά η Europol ε, θα λογοδοτεί και θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δημοκρατικό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι συμμετέχουν εδώ και τα εθνικά κοινοβούλια. Κυρίω επειδή και τα ίδια πρέπει να ελέγξουν τι ε, πληροφορίε στέλνουν οι εθνικέ αστυνομικέ αρχέ στην Europol, αλλά θα πρέπει να ελέγχουν και τι εκτελεστικέ αποφάσει που ε, λαμβάνει η αστυνομία και οι κυβερνητικέ αρχέ βάσει πληροφοριών που έχει λάβει από την Europol. Επιπλέον, τα εθνικά κοινοβούλια ε, θα πρέπει να προβαίνουν σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών και με άλλα κράτη-μέλη για να βλέπουμε ακριβώς πώς ε, λειτουργούν οι αστυνομικέ αρχές και οι μυστικές υπηρεσίες. Και θα είναι σε πολύ καλή θέση να αξιολογήσουν και να ελέγξουν κατά πόσο ε, η λειτουργία και ο κανονισμός της Europol συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Να μην δηλαδή αναλάβει ε, το έργο των εθνικών σας ε, αστυνομικών αρχών, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας. Έχουμε ακούσει τα όσα πρότεινε η Τρόικα, δηλαδή 62 άτομα που θα συνεδριάζουν ε, άπαξ ετησίως για 2-3 μέρες ενδεχομένως, για να δούμε πώς αυτό συνδέεται με την ανεξάρτητη εποπτεία των αστυνομικών αρχών, των μυστικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Αν δούμε την εντολή των περισσότερων επιτροπών σε εθνικό επίπεδο, κυρίως εστιάζονται στις ε, πολιτικές ε, της αστυνομίας της χώρας τους, των μυστικών υπηρεσιών, του υπερπολογισμού και της νομοθεσίας. Και επίσης ελέγχουν κατά πόσο η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες ε, συμμορφούνται με το κράτος δικαίου. Σε πολλές χώρες αυτοί οι φορείς λαμβάνουν και καταγγελίες για παράδειγμα πολιτών, αν θεωρούν ότι πλήττονται από την αστυνομία ή από τις μυστικέ υπηρεσίε. Κατά μέσο όρο, αυτοί οι κοινοβουλευτικοί φορείς έχουν από 5 έως 10 μέλη. Υπάρχουν και οι δεκιμάνσει, αλλά αυτό είναι ο μέσο όρο. Ποια είναι η σύνθεσή του. Συνήθω ε, τα μέλη έχουν ένα επαγγελματικό υπόβαθρο που συνδέεται, που άπτεται των αρμοδιοτήτων, αλλά όχι πάντα. Τουλάχιστον όμω κάτι πρέπει να ξέρουν για το τι ακριβώ ε, θα επιβλέπουν. Και για λόγους ε, δημοκρατική νομοποίηση είναι πολύ σημαντικό και τα πολιτικά κόμματα να εκπροσωπούνται σε αυτού του φορεί. Χωρί καμία εξαίρεση όλοι αυτοί οι φορεί έχουν και ε, προσωπικό 5-10 μελών και υπάρχει, υπάρχουν και εμπειρογνώμονες και διοικητικό προσωπικό. Εμπειρογνώμονες λοιπόν που έχουν λάβει επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. Σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά και σε χώρε όπω η Νορβηγία μπορούν να απευθυνθούν σε πυρογνώμονε κατά περίπτωση. Δηλαδή αυτοί οι εμπειρογνώμονε δεν συμμετέχουν ε, ε, στο προσωπικό, αλλά μπορεί η Επιτροπή να απευθυνθεί σε εκείνου όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Η συχνότητα των συνεδριάσεων. Και εδώ υπάρχει ποικιλομορφία, διαφέρει από το κράτο μέλο, αλλά μία φορά το μήνα, όπω στη Γερμανία, δύο φορέ το μήνα. Εξαρτάται και από το κάθε πότε, ε, κάθε πόσο συνεδριάζει και το ίδιο το κοινοβούλιο. Αυτό βλέπουμε πολλές φορές. Ε, σε πολλές χώρες ε, γίνονται και κλεισμένο των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις, γιατί δεν θέλουν να δώσουν μεγάλη, να τραβήξουν μάλλον τα φώτα της δημοσιότητας, Αυτέ οι δραστηριότητε δηλαδή να γίνονται πέρα από τα φώτα τη δημοσιότητα. όμως ε, οι εκθέσεις ε, που προκύπτουν είναι δημόσιες και μπορούν ε, κατά εξαίρεση να αποφασίσουν ότι μία συνεδρίαση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Πολλέ επιτροπές επίσης αποφασίζουν την κατανομή των αρμοδιοτήτων, ότι υπάρχουν δηλαδή υποεπιτροπέ ή ειδικοί σε ανά θέμα. Και το τελευταίο είναι η πρόσβαση στην πληροφορία. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ε, πληροφορίες. Στα περισσότερα κράτη-μέλη, ε, χωρίς ε, περαιτέρω αδειοδότηση, μόνο σε μερικά κράτη-μέλη αποφασίζεται οι βουλευτές να περνούν από μια διαδικασία ελέγχου. Οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες χάρη και μόνο στη θητεία τους. Δεν ισχύει το ίδιο για το προσωπικό. Εκείνοι ακολουθούν την συνήθη διαδικασία ε, ελέγχου υποβάθρου. Οργανώνονται ακροάσεις, έρευνες, επισκέψεις ε, στις ε, εγκαταστάσεις των υπηρεσιών που επιβλέπουν. Συναντιούνται με την ηγεσία της διοίκησης, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο και εκπονούν ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις. Κλείνοντας εδώ, μπορώ να πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ε, εθνικό επίπεδο, αν αποφασίσετε ότι αυτό θα είναι μια ε, καλή οντότητα, αν, αν το θέλετε, μπορώ να σας δώσω τις εξής συμβουλές. Όσο γίνεται λιγότερο, λιγότερα μέλη, και το 62 είναι αρκετά υψηλός αριθμός. Γίνεται ένα μήνυ κοινοβούλιο εντό εισαγωγικών. Μετά, αν συνεδριάζει μόνο μία φορά το χρόνο, με 62 μέλη και παραπάνω, τότε αυτό δεν λέγεται ελεγκτικός φορέας, είναι πλέον ε, συνδιάσκεψη. Αυτό είναι το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω. Ε, τρίτον, μεγαλύτερη συχνότητα συνεδριάσεων, αλλά και μεταξύ των συνεδριάσεων θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός υποεπιτροπών και εισηγητών με εξειδίκευση εξειδίκευση σε αυτά τα ζητήματα που θεωρείτε ότι χρειάζεται πιο εντελεχής ε, εξέταση. Μετανάστευση, οργανωμένο έγκλημα, γειτονικέ ε, δυνάμεις ε, που διασυνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα σας. Αν θέλετε λοιπόν να τα επιβλέπετε όλα αυτά, χρειάζεται ένα οργανωμένο σύστημα και μηχανισμός εισηγητών. Συμπερασματικά, Τώρα θα θεσπίσετε τον ιστορικό κανονισμό. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει να δούμε, είναι πολύ σημαντικό το τι μορφή θα λάβει αυτός ο ιστορικό κανονισμός. Και αν επιλέξετε υψηλότερο αριθμό μελών και χαμηλότερη συχνότητα συνεδριάσεων, θεωρώ ότι θα πρέπει ο ιστορικός αυτός κανονισμός να είναι όσο δυνατόν πιο ε, σταθερός, ε, να το έχετε καταλήξει και να υπάρχει και αυτός ο μηχανισμός μεταξύ των ε, συνεδριάσεων. Και περιμένουμε ενδιαφέρον να δω τα αποτελέσματα των εργασιών σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικός ομιλητής, πριν δώσουμε το λόγο στα μέλη, είναι Στρίνια Ρινίτσης. Από... η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας από το Κοινοβούλιο της Κροατίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα και μπορώ να σας μιλήσω για την πείρα μας από το Κοινοβούλιο της Κροατίας για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο προηγούμενος ε, μιλητής μίλησε πολύ καλά για την κατάσταση στην ε, Κροατία σε σχέση με αυτή τη θεώρηση πραγμάτων. Τη στιγμή που εγκρίθηκε το Σύνταγμα της Κροατίας έχουμε ε, ορίσει την ομοθεσία μας που κινείται με βάση τρεις πυλώνες. Και οι τρεις πυλώνες αυτοί διέπονται από το ε, Σύνταγμα και φυσικά υπάρχει και ένα σύστημα ελέγχων που ορίζει τη λειτουργία της όλης λειτουργίας. Προσπαθούμε λοιπόν να ελέγξουμε και να είμαστε υπόλογοι στο Σύνταγμα και φυσικά ως κυβέρνηση είμαστε ε, υπεύθυνοι για την εργασία μας και λογοδοτούμε. Μας απασχόλησε λοιπόν η εποπτεία των κυβερνήσεων και των Υπουργείων και αυτό αφορά και τις αστυνομικές δραστηριότητες και την αστυνομική επιθεώρηση. Υπάρχουν ειδικέ επιτροπές διερεύνησης εκεί όπου αρμόζει και με στα πλαίσια της ε, χορήγησης ψήφου εμπιστοσύνης είτε σε ολόκληρη την κυβέρνηση είτε στα επιμέρους χαρτοφυλάκια. Αυτά είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Οι πολίτες επίσης θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ετήσια λογοδοσία του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων για την δραστηριότητα της αστυνομίας και με βάση τα ερωτήματα των πολιτών. Πώς διενεργείται αυτή η κοινοβουλευτική έρευνα και εποπτεία. Λαμβάνουμε υπόψη όλες τη, ολόκληρη τη δραστηριότητα των αστυνομικών αρχών και αυτό γίνεται μέσω Υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπόλογο για τις δραστηριότητες της αστυνομίας και αυτό μετά το 1991 όταν συντάχθηκε το σύνταγμά μας. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ε, διενεργείται εποπτεία και έλεγχος από τις κοινοβουλευτικές αρχές χωρίς συζήτηση το 2000 το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο να λογοδοτεί κάθε δύο χρόνια στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κροατίας, γραπτός για όλες τις δραστηριότητες των αστυνομικών αρχών. Και αυτό να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά το δυνατόν. Μετά το 2011, με το νέο νόμο, υπάρχει μία ετήσια λογοδοσία, δηλαδή μία γραπτή διαδικασία, που αποστέλλεται στην Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά με βάση τους κανόνες υπάρχει, ε, και με βάση το Σύνταγμα υπάρχει η επίβλεψη των δραστηριοτήτων των αστυνομικών αρχών μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα. Και ο Υπουργός Εσωτερικών ετήσια υποβάλλει μία έκθεση για το προηγούμενο έτος και οι αστυνομικές αρχές, η αστυνομική διεύθυνση ελέγχεται από την, ε, από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά όχι, από, όχι άμεσα από τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά από έναν εκπρόσωπό του. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά το Υπουργείο Εσωτερικών να αποδίδει λογαριασμό στο Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή λοιπόν Εσωτερικών Υποθέσεων συζητά την έκθεση ετησίως. Στη συνέχεια εγκρίνεται ή απορρίπτεται και αποστέλλονται τα συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποδοχή ή μη της έκθεσης. Γι' αυτό υπάρχει μια ετήσια εποπτεία των ε, αστυνομικών αρχών. Βασιζόμαστε επίσης και στις αναφορές των πολιτών που υποβάλλονται έμεσα ή άμεσα. Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας βασίζεται και στις αναφορές των πολιτών σε σχέση με ενδεχόμενες παρατυπίες κατά τη δραστηριότητα των αστυνομικών αρχών κατά φυσικών ή νομικών προσώπων. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις αναφορές από άλλα ε, πρόσωπα τη στιγμή που υπάρχουν παρατυπίες. Υπάρχουν και οι ανώνυμες αναφορές, οι οποίες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών τη στιγμή που οι πολίτες δεν θέλουν να διαβιβάσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατά την προηγούμενη θητεία μας, μέσα στα πλαίσια ενός εξαμήνου είχαμε λάβει 31 αναφορές από πολίτες και τον τελευταίο μήνα το Κροατικό Κοινοβούλιο άρχισε να εξετάζει ε, εννέα παρόμοιες αναφορές. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναφοράς, ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί άμεσα ή έμεσα. Επίσης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών να ελέγξει όλες τις δηλώσεις αυτής της αναφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναφορά είναι τόσο περίπλοκη ώστε να χρειάζεται έλεγχος και από άλλους φορείς. Δηλαδή από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ή του Οργανισμού Καταπολέμησης της ε, Απάτης. Όταν ε, ληφθεί η αναφορά ε, συγκρίνονται τα στοιχεία με βάση την ε, απόφαση και την απάντηση του Υπουργείου και αποστέλλεται η απάντηση στον αναφερόμενο. Πολλές φορές αυτή είναι η τελική διαδικασία και συνήθως ο αναφέρον ικανοποιείται. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης μπορεί να γίνει επιπλέον έλεγχος από άλλους φορείς που εποπτεύουν τις αστυνομικές αρχές, όπως τον δημόσιο συνήγορο ή τον διαμεσολαβητή. Πολλές φορές οι αναφέροντες μας δίνουν νέα στοιχεία στην απάντησή τους και η Επιτροπή ζητά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι σχετικά χρονοβόρα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ικανοποιηθούν οι αναφέροντες. Η Επιτροπή επίσης μπορεί να προβεί σε έμεση εποπτεία ή έλεγχο και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αυτή προωθείται όταν υπάρχει και δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά και πολιτικό, σε σχέση με ενδεχόμενες παρατυπίες. Για παράδειγμα, έγινε ένας έμεσος έλεγχος με βάση αναφορές όταν έγινε λόγος για παράνομες δραστηριότητες κατά φυσικών προσώπων τότε ορίζεται μία ομάδα εργασίας και ε, πραγματοποιούνται και επισκέψεις εκεί όπου επιβάλλεται. Και γίνονται και συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους. Με βάση την τεκμηρίωση, το περιεχόμενο αυτών των συνεντεύξεων ή τα αποδεικτικά στοιχεία οδηγούν σε αποφάσεις για το κατά πόσο υπήρξε παραβίαση του νόμου και σε τέτοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το κατά πόσο ο αναφέρον είναι ή ικανοποιημένος ή μη, ε, αποστέλλεται απάντηση στον, στον αναφέροντα. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία και εάν γίνει απαγγελία κατηγοριών τότε εμπλέκεται και ο δημόσιος κατήγορος. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή εσωτερικών υποθέσεων ασχολείται εκ του σύνεγγης με τέτοιες ε, περιπτώσεις και όχι μόνο με αναφορές αλλά και με άλλες δραστηριότητες αν και πιστεύει ότι οι αναφορές είναι πολύ χρήσιμες. Επίσης άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν με βάση τις αναφορές από τους πολίτες. Πολύ συχνά οι αναφέροντες κάνουν λόγο για παρατυπίες στην δραστηριότητα της αστυνομίας, των αστυνομικών αρχών, έτσι ώστε να υπάρχει εκ του σύνεγγης έλεγχος πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για όλη την ε, υπομονή σας. Παλιότερα μοιράζαμε καφέ για να ξυπνάτε, αλλά τώρα ε, κάνουμε οικονομίε, αλλά υπάρχει έξω ένα μηχάνημα με καφέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σας ενθαρρύνω να βγείτε, αλλά έχετε υπόψη σα ότι υπάρχει ένα μηχάνημα που πουλάει καφέ. Αν θέλετε καφέ, παρακαλώ. Είναι Δευτέρα απόγευμα. Τώρα να αρχίσουμε απευθεία τη συζήτηση. Έχουμε, θα έχουμε την αναθεωρημένη πρόταση μέσα Δεκεμβρίου και η τελική πρόταση Μάρτιο ή Απρίλιο. Πότε είπατε? Μάρτιο ή Απρίλιο, μάλιστα. Οπότε θέλουμε να μα πείτε τώρα πώς θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της πρότασης και τι άλλα σχόλια έχετε. Λοιπόν και πάλι παρακαλώ δύο λεπτά, ε, δύο λεπτά. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Οκέιλεν από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχω μια σειρά από για την πρόταση αυτή. Πώς ακριβώς θα εκπροσωπούνται τα εθνικά κοινοβούλια. Εδώ λέει με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Δύο αν κοινοβούλιο και αν έχουμε δύο νομοθετικά σώματα σε μια χώρα, ένα από κάθε νομοθετικό σώμα. Αλλά δεν καθορίζει πώς θα καθοριστούν τους, οι έξι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς λοιπόν θα επιλεγούν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, συχνότητα συνεδριάσεων. Στη γενική παρουσίαση για τη σημερινή μας συνεδρίαση τονίζεται ότι η Europol πρέπει να είναι υποσωστό σωστό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η λέξη σωστός είναι πολύ σημαντική. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι σημαίνει. Βεβαίω, δημοκρατικό έλεγχο, αλλά σωστό είναι όντω σωστή η διαδικασία ελέγχου με έναν, με συγγνώμη, με μία συνεδρίαση το χρόνο. Τι σημαίνει λοιπόν. Απλώς θα αντιδρούμε σε μία ετήσια έκθεση. Δεν θα μπορούμε να παρέμβουμε απευθείας για να ελέγξουμε την Europol και τις ε, διάφορες διαδικασίες της. Θα ήθελα να μου πείτε πώς νομίζετε ότι θα ενημερώνονται σωστά τα μέλη της ομάδας αυτής για τις εξελίξεις και την ε, δραστηριότητα της Europol και πώς αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να ληφθεί σωστά υπόψη και πώς θα καθορίζουμε εάν χρειαζόμαστε μια δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση κατά κάποιο ημερολογιακό έτος. Ευχαριστώ κύριο Κίλεν. Σας ευχαριστώ πολύ σωστές ερωτήσεις σας. Ο κύριος Χάμερμπεργκ από τη Σουηδία. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλοί είπαν ότι η συνεργασία αυτή είναι απολύτως αναγκαία το κυβερνοέγκλημα, ξέρετε, κάθε τρει μήνες διπλασιάζεται. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι απόλυτα απαραίτητη και η δραστηριότητα των εθνικών και τοπικών αρχών. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος λοιπόν, αλλά πρέπει να είναι ουσιώδης. Δεν θα πρέπει απλώς να τα λέμε που και που. Θα πρέπει να πιστεύουν όλοι ότι η Επιτροπή αυτή, η ομάδα αυτή κάνει σωστή δουλειά. Βεβαίω πρέπει να έχουμε εκπροσώπου από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτοί ξέρουν πώ λειτουργούν οι τοπικέ και εθνικέ αστυνομικέ αρχέ. Τίποτα δεν μας εγγυάται ότι μια νέα γραμματεία και νέες δαπάνες σημαίνουν περισσότερη αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι αν αξιοποιήσουμε τους σωστούς κοινοβουλευτικούς μπορούμε να ασκήσουμε ουσιώδη έλεγχο χωρίς νέες δομές. Ο συμβασμός νομίζω ότι είναι καλός. Δεν πρέπει να είμαστε διαστάσεις, να έχουμε διαστάσεις κοινοβουλίου. Δύο με τρεις από κάθε κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι ο σωστός αριθμός και μια δυο συνεδριάσει το χρόνο. Και αυτό νομίζω είναι καλό. Αλλά όσο Σουηδοί μας ανησυχεί λιγάκι όλη αυτή η συζήτηση για νέε δομέ, νέα σώματα, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές τι θα κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και αυτό είναι ιδιαίτερα καλό. Ο κύριο Πέρεθ Λαπαθεράν από την Ισπανία. Ευχαριστώ. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες ε, που δεν απάντησε στο ε, ερωτηματολόγιο γιατί επίκεντρο εκλογές και χρειάστηκε να περιμένουμε. Είχαμε δύο εκλογές ε, πολύ κοντά τη μία στην άλλη. Τώρα όμως υπάρχει περισσότερη πολιτική σταθερότητα, δεν είναι προσωρινή η κατάσταση και θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση για να απαντήσουμε σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι δεν αρκεί μία συνεδρίαση το χρόνο. Για να υπάρχει εμπλοκή χρειάζεται περισσότερες ε, συνεδριάσεις, τουλάχιστον δύο το χρόνο. Γιατί έτσι θα ασκήσουμε καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αριθμός μελών. Και ιδίω ε, σε κάποιες χώρες που έχουν δύο νομοθετικά σώματα, έτσι μπορούμε να ε, ε, ε, υπάρχει περισσότερη εκπροσώπηση των διαφόρων ε, τάσεων και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν δύο. Δύο από τη Βουλή και δύο από τη Γερουσία. Ο κύριος Ντεμέρα λέει να είναι ευέλικτο το όργανο, αλλά θα μπορούσε κάθε χώρα να έχει ένας-δύο εκπροσώπους, για παράδειγμα, για τις συνεδριάσεις. Έτσι θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα καθήκοντα. Επίσης θεωρούμε ότι θα τα πάμε καλύτερα. Θέλουμε ένα όργανο κοινωνικού ελέγχου. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα διαχειριστικό όργανο. Θέλουμε απλώς να συλλέγουμε πληροφορίες και να κυκλοφορούν προτάσεις. Δύο συνεδρία στον χρόνο, με τέσσερι εκπροσώπους ανά χώρα. Και για την Προεδρία, ναι. Μπορούμε να εγκρίνουμε την πρόταση, μια συμπροεδρία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της εναλλασσόμενης ε, Προεδρίας της Ένωσης. Ε, δύο συνεδριάσεις το χρόνο είναι ακριβώς όπως γίνεται και με τις Προεδρίες της Ένωσης, που είναι δύο το χρόνο. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόταση, ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της χώρας μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Γερμανία και Χάκμαν. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντίαθ Δεμέρα, ο οποίος ε, για πολλά χρόνια και με διάφορες αρμοδιότητες προώθησε αυτό το θέμα με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, με πολλή δέσμευση και νομίζω ότι όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε και άλλους βέβαια, αλλά ιδίω εκείνων για αυτά που επετέχθησαν. Κάτι που είναι απόλυτα σαφές από όλες τις παρουσιάσεις. Η Europol χρειάζεται περισσότερες αρμοδιότητες. Πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Αλλά η Europol πρέπει να μπορέσει να εργαστεί. Αλλά παράλληλα Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Το τονίσατε. Εμπιστοσύνη προς την Europol θα υπάρχει μόνο εάν αυτές οι επιπλέον αρμοδιότητες ε, όπως σε τα δοχεία συμπληρώνονται από συμπληρωματικού και αποτελεσματικού ελέγχου. Αυτή είναι η σωστή ιδέα. Και εμεί την υποστηρίζουμε βεβαίω ω Γερμανία. Η Γερμανική Βουλή ε, υπέβαλε αναλυτικές προτάσεις και καταλήγουμε ότι για μια σειρά θέματα πρέπει ακόμη να διευκρινιστεί η κατάσταση. Μέσα Δεκεμβρίου το αποτέλεσμα της συνάντησής μας θα το έχουμε. Αλλά δεν είναι η τελική φάση της εργασίας μας. Προτείνουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα με βάση τις διάφορες προτάσεις να συναντηθούμε άλλη μια φορά για να τα εκτιμήσουμε όλα αυτά και να τα, να τα συνδυάσουμε. Για παράδειγμα, ε, το θέμα των ε, δικαιωμάτων της μειοψηφίας είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θεωρούμε ότι κατά τη γνώμη μας χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις αναχώρα. Γιατί βεβαίω αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα πρέπει να έχουμε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει και αντιπροσωπευτικότητα. Και αν η αντιπροσωπευτικότητα δεν είναι επαρκής τότε το σώμα αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό. Δεν θα το παίρνουν σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση για τέσσερις αναχώρα και επιπλέον θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθεί πριν αρχίσει να λειτουργεί το σώμα τρόπος για να καθορίσουμε πώς θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των μειοψηφιών, πώς θα οργανωθεί το σώμα, τι στοιχεία θα λαμβάνει και τελευταία παρατήρηση, τα θέματα της αστυνομίας είναι βεβαίως ευρωπαϊκά αλλά σε μεγάλο βαθμό ακόμη εθνικά θέματα. Γι' αυτό είναι καλό να υπάρχει η σωστή και ισότιμη εκπροσώπηση. Ευχαριστώ την τελεία κύριε Λαμόρο. Συνάδελφοι, ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη Λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αφορά κοινέ ευθύνε των ε, κοινοβουλίων. Εμείς ε, μπορούμε να ελέγξουμε την ε, τήρηση των δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών στα πλαίσια άσκησης της ε, πολιτικής ασφάλειας. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να υπάρχει ένας κοινό ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος για να δημιουργήσουμε ένα κοινό τόπο περί μετά από 7 χρόνια, μετά δηλαδή τη θέση εφαρμογή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε λοιπόν ότι η Τρόικα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να ασκήσει σωστά αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ε, δρούμε με βάση το απόρριτο, αλλά να υπάρχει πραγματικός πολιτικός έλεγχος και εποπτεία με βάση τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ. Και για αυτούς τους λόγους ακριβώς και με βάση και την ε, προγενέστερη παρέμβαση θα ήθελα να προτείνω για κάθε κοινοβούλιο να γίνει μια αυστηρή επιλογή για την ε, εξειδικευμένη αυτή επιτροπή για να υπάρχει μια συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Ο αριθμός ε, λοιπόν των βουλευτών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένος έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικός πολιτικός έλεγχος ε, της Ευρωπόλ με βάση υποομάδες που ακολουθούν, παρακολουθούν συγκεκριμένες θεματικές όπως την εγκληματικότητα και να συνέρχονται μία φορά το χρόνο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να, προβλέπονται, να προβλέπεται και η δυνατότητα έκτακτων ε, συνεδριάσεων καθώς και ένα σημείο επαφής για να γίνει μία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Από το Λουξεμβούργο, ο κύριος Άγγελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τους συναδέλφους που συμμετείχαν ε, στην ομάδα εργασία κυρίως ε, τη συνάδελφα από την Σλοβακία και τον κύριο Δίας Δεμέρα, εκπρόσωπο του Ευρωκοινοβουλίου και μεγαλογνώστη του ζητήματος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ε, το πνεύμα συνεργασίας που υπήρχε σε αυτήν την ομάδα εργασίας και υπενθυμίζω ότι οι εργασίες... Ε, συνάδουν πλήρω με τον βαθμιδόν αυτόν οδικό χάρτη που αποφασίστηκε το 2016 το Μάιο Αν δούμε τι απαντήσει του ερωτηματολογίου, συμπεραίνουμε ότι όλοι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό και να βρούμε λογικέ λύσει. Και αναμφίβολα, κοινό στόχο είναι να έχουμε έναν αποτελεσματικό, μικρό και εξειδικευμένο ε, μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όλοι ξέρουμε ότι είναι η ευθύνη μα να παρακολουθούμε από πολιτική σκοπιά στι ε, δραστηριότητε ε, τη Europol, σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι ελευθερίε. Γι' αυτό έχουμε καθήκον προ του πολίτε να έχουμε έναν ε, μηχανισμό, έναν φορέα ευέλικτο και αποτελεσματικό και όχι ένα μεγάλο φόρουμ συζήτηση. Συζητούμε σήμερα τις βασικές λεπτομέρειες όπως είναι η σύνθεση ε, της ομάδας, ε, ο τόπος εξαγωγής ε, των δραστηριοτήτων και ούτω καθεξής. Ήδη όλα αυτά είναι αρκετά πολύπλοκα από μόνα τους, γι' αυτό υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή και καθήκον μας, η εντολή μας δηλαδή, υπάρχει στο άρθρο 51 του νέου κανονισμού ε, της Europol. Τα υπόλοιπα πρακτικά ζητήματα λοιπόν που έχουν θίξει οι συνάδελφοι θα πρέπει ε, να τα διαχειριστεί η ίδια ομάδα. Ζητήματα γραμματείας, εμπιστευτικότητας κτλ. Η ίδια η ομάδα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει αυτά τα ζητήματα. Και στο παρελθόν με άλλους τέτοιους ε, διακοινοβουλευτικούς φορείς ε, ε, απεδείχθη δύσκολο να εξευρεθεί ε, συνένεση για, αυτό, για τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά θα συμφωνήσουμε πρώτα για αυτό το βήμα, να συνέλθει η ομάδα των σημαντικών δυνατών. Έχουμε τον οδικό χάρτη που μας εξήγησε η μιλήτρια προηγουμένως. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει με βάση αυτόν τον οδικό χάρτη να κινηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα, ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Μπόρν που εκπροσωπούσε ε, το κέντρο από τη Γενέβη. Γιατί με ενδιαφέρει αυτή η συγκριτική ανάλυση για τα, τις διάφορες μορφές των μονάδων που έχουν σχέση ε, με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και αυτές τις μελέτες για την αστυνομική συνεργασία και μιλήσατε για τη συμμετοχή, ε, τη διάρκεια της εντολής, την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων ομάδων, όμως στη σύγκριση αυτή δεν υπήρχε ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ σημαντικό. το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και πιο συγκεκριμένα ποιε είναι οι κυρώσει που προβλέπονται, ποιε είναι οι πολιτικές προεκτάσεις και συνέπειε ε, για να υπάρχει πραγματική πολιτική ε, λογοδοσία και να απαιτούμε την πολιτική ευθύνη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για μια συγκριτική ανάλυση, λαμβάνοντα υπόψη ότι στα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια ο κοινοβουλευτικό έλεγχο οδηγεί στην ε, απόδοση κοινοβουλευτικών ε, ευθυνών και αυτό μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να οδηγεί ακόμα και σε παρετήσεις των επικεφαλής ε, ορισμένων επιχειρήσεων που δεν ε, κατάφεραν ε, να αποκομίσουν την ε, έγκριση του Κοινοβουλίου και αυτό βέβαια συμβαίνει σπάνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των επιχειρήσεων της Europol, ποια είναι η δική σας νόμη. Ευχαριστώ. Επανέλθ, επανέρχομαι στους υπουργούς των Δικοκοινοβουλίων, ο κύριος Σόλη. Ευχαριστώ. Αρχικά να γνωρίζω ε, και χαίρομαι για την αναγνώριση μάλλον που έλαβε η Βουλή των Λόρδων για τα όσα έχει κάνει και μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει και άλλη έκθεση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλεία και υπό το φω ε, του Brexit. Θα το δημοσιοποιήσουμε αρχής γενομένης από τις 12 Δεκεμβρίου. Νομίζω και εγώ ότι είναι πολλά τα 62 μέλη για το κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά λαμβάνοντα υπόψη όλε τι ομάδε και πολιτικά κόμματα θα πρέπει να εκπροσωπηθούν, μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, δεδομένων των συνθήκων. Αυτό που με προβληματίζει τώρα είναι η συχνότητα των συνεδριάσεων. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μπόρν έχει δίκιο όταν λέει ότι θα είναι περισσότερο μια συνδιάσκεψη, ε, τρει μέρε μια φορά το χρόνο ας ξεκινήσουμε με δύο συναντήσεις ε, το χρόνο και να το επανεξετάσουμε. Και αυτό το λέω για δύο λόγους. Είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο όταν έχουμε ε, συνεδριάσει σε ανατακτά χρονικά διαστήματα και κατά δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, εξετάζονται ζητήματα δικαιοσύνης δεν θέλουμε μόνο την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και την πραγματική της απόδοση. Πώς δηλαδή θα διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό ισχύει ευρύτερα. Ε, και στο πλαίσιο μια χώρα ε, που έχει επιλέξει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να το πω αυτό. Και ένα από του λόγου που έγινε αυτό ήταν ε, αυτή η αίσθηση τη έλλειψη λογοδοσίας από πολλού φορεί. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Η προβολή και ορατότητα ενό τέτοιου φορέα μπορεί να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποστείλει το μήνυμα ότι τα εκλεγμένα μέλη των κοινοβουλίων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεριμνούν για την ε, λογοδοσία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Υποδεχόμαστε λοιπόν, και τον κύριο Κούπερ που ε, τώρα από, από εδώ και πέρα συμμετέχει στην ε, σχετική αρμόδια επιτροπή στη χώρα μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Nordquest από τη Δανία, παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, στη Δανία δεν ξέρουμε ακριβώς ε, πώς ε, θα συνδεθούμε με την Europol, όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, γιατί τα δεδομένα, οι πληροφορίες είναι εξουσία και ισχύς. Και είναι σημαντικό όταν ε, δίνουμε τέτοιες εξουσίες στην Europol, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και ο σχετικός έλεγχος. Είναι πολύ καλή πρόταση που έχει υποβληθεί. Πρέπει να δούμε τώρα για τον αριθμό των μελών. Εντάξει, θα το δούμε. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο τρόπος λειτουργίας Πώς λοιπόν θα εξετάζει συγκεκριμένε υποθέσεις μια τέτοια ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, αν θα υπάρχει δυνατότητα για τους ίδιους τους πολίτες ε, να το πράξουν. Μπορούμε να εξετάσουμε και τις πρακτικές λεπτομέρειες, πόσο θα είναι το χρόνο κτλ. Όμως το πιο σημαντικό είναι το περιεχόμενο ε, της λειτουργίας. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πρώτα και κύρια. Πώς θέλουμε ακριβώς να επιτελείται αυτό το έργο αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Με εξέπληξε η συντομία του σχολείου σας. Τώρα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριο Τερικάπρας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολλά και ενδιαφέροντα ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Τέσσερα είναι τα σημεία που είναι σημαντικά για μια σωστή εποπτεία από την ε, μεικτή ομάδα. Οι μειοψηφίες, ε, οι κοινοβουλευτικές μειοψηφίες θα πρέπει να εκπροσωπούνται στη νέα ομάδα, μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικής εποπτείας για να εισακουστεί η φωνή τους. Αυτό έχει σχέση και με τη σύνθεση της ομάδας, τη διαδικασία ψηφοφορίας, απαρτία, ε, ορισμός ε, επιτροπών διερεύνησης και ούτω καθεξής. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία για όλα τα κοινοβούλια και βουλευτές. Τρίτον, ο έλεγχος θα πρέπει να οδηγήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, να είμαστε κοντά στους πολίτες με δημόσιες ακροάσεις. Ίσως θα πρέπει να συμμετέχει και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τέταρτον, μία ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο σώμα. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικό στην εργασία του. Επειδή πολλά κράτη-μέλη έχουν ένα μόνο ε, κοινοβουλευτικό σώμα, θα μπορούσαμε να έχουμε μία συνάντηση ετησίως που να, που να διαρκεί δύο ημέρες. Ξέρω ότι αυτό που θα πω ίσως αντιτίθεται στην πλειοψηφία, αλλά θα πρέπει να πω την προσωπική μου άποψη. τα μέλη θα πρέπει να είναι 30 κατά το μέγιστο, ένα για, ένα για κάθε κράτος μέλος και έξι βουλευτές, δηλαδή ο εισηγητής και οι σκιώδης που εργάζονται για τον κανονισμό που συντάσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στάουτς από την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πεπισμένοι στην Ουγγαρία ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις και η απειλή της τρομοκρατίας είναι κάτι το πολύ απτό και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία της Ευρωπόλ για το, ε, για το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η τρομοκρατία πολλές φορές συνδέεται με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα μέσω αυτής της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου θα μπορέσουμε να πλήξουμε και τους ενδυνάμει τρομοκράτες κατά αυτόν τον τρόπο. Θα συλλέξουμε πληροφορίες αλλά και θα τις αναλύσουμε. Στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες στα κράτη-μέλη και έτσι μπορούμε να δράσουμε από κοινού. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι ύψης της σημασίας. Σίγουρα θα επιτελεστεί πρόοδος. Τι θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι μία ετήσια συνάντηση δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε δύο συναντήσεις ετησίως για να είναι αποδοτικός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και ίσως δεν αρκούν ούτε αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία εκπεριτροπής προεδρία η οποία και να φιλοξενεί αυτές τις συναντήσεις ως προς το γλωσσικό καθεστώς το άρθρο 7 των κατευθυντηρίων γραμμών της Στοκχόλμης θα πρέπει να ισχύσει, όπως ισχύει και για τη διάσκεψη των ε, Προέδρων. Ευχαριστώ. Δημητρίου από την Κύπρο. Ε, εμείς ως Κύπρος θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι προτεραιότητες που θα έχει αυτή η μειχτή κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα επιτελεί τον ρόλο του ο αριθμός, όπως έχει πει και ο κύριος Τίας Δεμάρε και ο κύριος Μπορ, είναι πολύ σημαντικό να είναι τόσος που να είναι ευέλικτο το σώμα. Δεδομένου το όσα ακούστησαν, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό με λιγότερους από δύο μέλη από κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο, συν τα έξι μέλη του Ευρωπαϊκού Βουλίου. Άρα πάμε αμέσως στα 62. Άρα, η συχνότητα των συνεδριάσεων σίγουρα πρέπει να είναι περισσότερες από μία, για να μπορεί ακριβώς αυτό το όργανο να μην έχει ρόλο διεκπαιρεωτή και να λειτουργεί, όπως πολύ σωστά το είπε ο κύριος Μπορ, ως σε συνδιάσκεψη. Ε, από εκεί και πέρα, η κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να έχει την ε, ευελιξία να επιλέγει η ίδια ποια θα είναι τα μέλη αυτά και τι εμπειρογνωμοσύνη ακριβώς θα έχουν. Τα μέλη να επιλέξουν την ε, σοβαρότητα που θέλουν να δώσουν σε αυτό το σώμα, σε αυτή τη μεικτή επιτροπή. Οι έκτακτες συνεδριάσεις θα πρέπει να είναι, δεν πρέπει να τελεί υπό τον αίρεση του Κοινοβουλίου του κράτους, μέλους, πρέπει να είναι δεδομένοι. Ε, αν θα δημιουργηθούν υποεπιτροπές, ακριβώς για να δοθεί έμφαση στον ρόλο αυτής της, υπο, της ε, επιτροπής, η εκπροσώπηση όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να διασφαλίζεται. Εάν οι εν λόγω σχηματισμοί θα έχουν επιλεκτικά ενισχυμένη η προνομιακή και άρα άνηση πρόσβαση σε πληροφορίες για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Η εμπιστευτικότητα θεωρούμε ότι είναι σαφές ότι θα τηρείται όπως τηρείται και στα εθνικά μας κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα έπρεπε να σας ε, αναφέρω ότι μεταδίδεται αυτή η συνεδρίαση στο διαδίκτυο. Γίνεται άμεση αναμετάδοση, κάτι το οποίο δεν προανέφερα. Ο κύριος Σεπάρας από την Λιθουανία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν σε πολλά σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αρκετά από αυτά. Σήμερα μιλάμε για μια διαφορετική μορφή δραστηριότητας όπου συνυπάρχουν Ευρωπαϊκό με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θέλουμε να επιτύχουμε γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προωθηθεί και στον τομέα της δικαιοσύνης μέσω Eurojust. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια και στα κράτη ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις ως προς το μέγεθος της ομάδας αυτής, αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα καθήκοντά της. Θα οργανώνει μόνο τις ακροάσεις ή θα ακολουθήσει τον τρόπο δραστηριότητας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπόλ και Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν επιλέγουμε τους εκπροσώπους, διότι η ομάδα θα ασχοληθεί με ευαίσθητες πληροφορίες και εμπιστευτικού χαρακτήρα. Γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη για το, ως προς το μέγεθος της ομάδας. Ο προλαλής σας είπε κάτι το πολύ σκόπιμο ότι θα μπορούσαμε και να λειτουργήσουμε υπομορφή ε, υποεπιτροπών. Έχουμε ακόμη δύο εκπροσώπους για, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επειδή όμως ε, πρέπει να φύγει η κυρία Φούνερ, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα. Είχατε πει ότι θα φεύγατε νωρίτερα. Θέλετε να αντιδράσετε τώρα και μετά θα είναι η κυρία Κοζομπόλη και ο κύριος Σερνόφσκι. Μετά και μετά θα πάρουν το λόγο οι ε, άλλοι ομιλητέ. Ευχαριστώ πολύ. Από μέρους μου και από πλευράς όλης της ομάδας εργασίας να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, την επικοδομητική σας ε, συμβολή και προτάσεις. Χαιρόμαστε που η δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα για τις λεπτομέρειες ε, της λειτουργίας ε, αυτής της ε, κοινή κοινοβουλευτικής ομάδας ελέγχου ε, αντιμετωπίστηκαν θετικά από πολλούς από τους ομιλήσαντες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περισσότεροι από ό,τι άκουσα στηρίζουν την, άποψη, την προσέγγιση μας. Βεβαίω, οι συζητήσει ε, επίση απέδειξαν ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσει. Η ομάδα εργασία, όπω ε, προείπα, θα επιχειρήσει τώρα να αναλύσει όλα τα σχόλια που ακούσαμε ήδη σήμερα και θα σας υποβάλει μια νέα πρόταση ε, μέχρι τις 16-12 του τρέχοντος. Σήμερα έχουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ακούσαμε πολλές συγκεκριμένες προτάσεις για την λειτουργία, τις λεπτομέρειες λειτουργίας αυτής της ομάδας. Ορισμένε θα μπορούσαν για παράδειγμα να μπουν σε έναν εσωτερικό κανονισμό αυτής της ομάδας. Όπως είπαμε και στην αρχή, ε, ε, στα πλαίσια τη εντολή τη, η ομάδα εργασίας κυρίως εστίασε στα βασικά θέματα λειτουργίας του σώματος ούτω ώστε να αποφασιστούν μέχρι τον Μάιο του 2017. Γιατί θέλουμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Να έχουν καθοριστεί μέχρι τότε οι βασικέ αρχέ λειτουργία. καθώς και οι κυριότερες, ε, οι βασικές λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας και τα περαιτέρω θέματα θα συνεχίσουν ε, να είναι υποσυζήτηση. Οτιδήποτε έχει συμφωνηθεί μέχρι τότε θα μπει σε αυτήν την επόμενη πρόταση που θα σας κάνω. Ευχαριστώ πολύ και χαίρετε. Οι συνεργάτες της, λέει ε, είναι ακόμα εδώ. Θα ακούσουμε άλλους δύο μιλητές και ούτως άλλως συνεχίζει τη διαδικασία όπως σας εξηγήσω προς το τέλος αλλά χαίρομαι που μπόρεσε να αντιδράσει έστω και μερικά πριν χρειαστεί να φύγει. Η κυρία Κοζομπόλη, παρακαλώ, από την Ελλάδα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικώς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ομάδα εργασίας και ιδιαίτερο στη Σλοβάκικη Προεδρία για την εργασία που κατέβαλε προκειμένου να διευκολύνει την δουλειά όλων μας. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια. Ως προς το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε, η Βουλή των Ελλήνων είναι σύμφωνη με αυτό που έχει προταθεί. Το προτινόμενο σχέδιο επιτυγχάνει μια ικανοποιητική ισορροπία στην εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων εξυπηρετεί τόσο τη διευκόλυνση ουσιαστικού διαλόγου και επαφών ανάμεσα στα μέλη του σώματος, όσο και τις υποχρεώσεις εχεμήθειας που συνεπάγεται η συμμετοχή στο κοινοβουλευτικό έργο. Αναφορικά όμως με το τρίτο θέμα θα έλεγα ότι η βούληση των περισσότερων κοινοβουλίων εκφράζεται ορθότερα από τη διοργάνωση της διάσκεψης δύο φορές το χρόνο και όχι μία. Αν δεν κάνω λάθος, 22 από τα σώματα που απάντησαν εκφράζουν την άποψη αυτή έναντι 10 που στηρίζουν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων μία φορά το έτος. Προκειμένου δεν να επιτύχουμε πάλι μια ικανοποιητική ισορροπία, θα πρότεινα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης κατά το πρώτο εξάμεινο στην Προεδρεύουσα χώρα και κατά το δεύτερο εξάμεινο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η δαπάνη οργάνωσης της κοινοβουλευτικής διάστασης τη Προεδρία για τα Κοινοβούλια του Θερινού Εξαμήνου που διοργανώνουν επιπρόσθετα την διάσκεψη Προέδρων, Γενικών Γραμματέων, ε, οικονομική διακυβέρνηση κτλ. Ενώ αξιοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ω προ την ουσία του πράγματο, οι διπλέ συνεδριάσει θα διευκολύνουν και το έργο των βουλευτών που καλούνται να ελέγξουν ένα μεγάλο όγκο εγγράφων και εκθέσεων, όπω προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού η μεικτή Επιτροπή του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου θα μπορούσε το πρώτο εξάμεινο να εξετάζει την έκθεση υπεπραγμένων του προηγούμενου έτους και να την αξιολογεί. Εδώ κατατίθεται ε, γίνεται μια έκκληση να κατατίθεται η έκθεση αυτή εντός του Ιουνίου εκάστου έτους ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες της Επιτροπής. Το δεύτερο εξάμεινο να εξετάζεται ο προγραμματισμός του επόμενου έτους με παρεμφερή τρόπο λειτουργεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, ε, η Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας. Δεδομένης της κρίσιμης συγκυρίας για τα ζητήματα ασφάλειας αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας των θεμάτων αστυνομικής συνεργασίας και του πλούσιου νομοθετικού έργου που σωστά προωθεί η Ευρωπαϊκή okay, Επιτροπή σε ζητήματα που αγγίζουν τα προσωπικά δεδομένα, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει έντονος okay, διάλογος και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Okay, thank you. We're, we're running out of time. Ευχαριστώ πολύ. Thanks. Mr. Δεν έχουμε χρόνο για αυτό σας διακόπτω. κύριο Σινόφσκι, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Τρόικα για αυτές τις προτάσεις και για το δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο τα εθνικά κοινοβούλια συμμετείχαν στην διαβούλευση. Και διαπιστώνουμε από αυτές τις προτάσεις ότι έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί συμβιβασμός. Η ε, ερώτηση 1 είναι αυτονόητη. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αποφασίζουν. Αυτοί ξέρουν ποιοι μεταξύ των μελών τους είναι οι πιο κατάλληλοι για ένα τέτοιο σώμα. Για τη δεύτερη ερώτηση για το θέμα δηλαδή του αριθμού εκπροσώπων από κάθε σώμα. Από τη μία βέβαια υπάρχει το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας, λειτουργικότητας ε, ενός ε, τέτοιου σώματος, αλλά από την άλλη επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι αν περιοριστούμε σε δύο μόνο μέλη ανά χώρα, δεν μπορούν να εκφραστούν οι διαφορετικές τάσεις που εκφράζονται διαφορετικέ τάσει των κοινοβουλίων. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση. Γι' αυτό προτείνουμε έξι εκπρόσωποι από κάθε κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποιες δυσχέρειες, αλλά ε, νομίζουμε ότι οι προτάσεις της Γερμανίας και της ε, ε Ισπανίας για τέσσερις είναι ικανοποιητικέ. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τρίτη ερώτηση. Συχνότητα συνεδριάσεων, τόπο συνεδριάσεων. Για μας αυτά είναι τα θέματα που μας δημιουργούν ε, τις περισσότερες δυσχέρειες. Αλλά ίσως θα υπήρχε δυνατότητα και εδώ να επιτευχθεί κάποιο συμβασμός. Πολλοί είπαν ότι δεν αρκεί μια συνεδρία στον χρόνο. Άρα μια λύση που θα μπορούσε να εξεταστεί και που τηρεί κάποιες αρχές που μας είναι ιδιαίτερα αγαπητές. Πάντα η Προεδρία διοργανώνει τέτοιου τύπου συνεδριάσεις κάθε Προεδρία και η δεύτερη συνεδρίαση γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή θα είχαμε τρει συνεδριάσεις το χρόνο. Δύο για κάθε Προεδρία, δηλαδή μία για κάθε Προεδρία αναξάμεινο και μία τρίτη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα πρώτος έχει το λόγο για να απαντήσει στι ερωτήσει που του έθεσαν συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα αντιδράσω πολύ, θα απαντήσω πολύ ε, τηλεγραφικά στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη συζήτηση αυτή. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνω μια αρχική διευκρίνηση. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να πω το εξής. Η Ευρωπόλ δεν είναι ένας οργανισμός που μπορεί να επιβάλλει αποφάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να συγκριθεί με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών. Εμείς αυτό που ελέγχουμε ή θα ελέγξουμε δεν είναι αστυνομικές αρχές ε, κρατών μελών. Πρόκειται για μία αρχή που δεν έχει, οι αποφάσεις οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να επιβάλλει τις αποφάσεις της. Η Ευρωπόλα αφορά τη συνεργασία, αφορά την ε, εξέταση των πληροφοριών και οι πληροφορίες, ε, επεξεργασία πληροφοριών μάλλον, που αφορούν την εγκληματική δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να βγάλετε από το νου σας αυτή τη δυνατότητα ελέγχου κρατικών αστυνομικών αρχών, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Μπόρν μας έδωσε πολλές πληροφορίες, εμπλούτησε τις γνώσεις μας σε σχέση με το δημοκρατικό έλεγχο των ενόπλων ε, δυνάμεων. Και μας εμπλουτίζει ακριβώς για το δημοκρατικό έλεγχο που μπορεί να ασκηθεί και σε άλλους ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Εμείς όμως μιλάμε για την Ευρωπόλ εδώ και τις δυνατότητες και τα όρια της. Τώρα, άλλες ερωτήσεις. Μία που με αφορά, με αφορά ως διαπραγματευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είπα ότι είμαι αλληλέγγυος με τις ε, προτάσεις συμβίβασμου της Τρόικας, αλλά δεν υπέρ του να υπάρχουν έξι εκπρόσωποι, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζει και ο πρόεδρος Μωράης, ελήφθη μία απόφαση του Συμβουλίου χωρίς όμως να υπάρχει μία ε, διάρθρωση η οποία προϋπάρχει. Δηλαδή, δεν θα δεχτεί κανείς ένας διαπραγματευτής να ορίσει και να σταθεί στους έξι. Και αυτό θα ήθελα να το τονίσω, να το θέσω επιτάπητος. Δηλαδή, η Τρόικα και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να δεχτούν μία σχετικά χαμηλή ή περιορισμένη εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι το άρθρο 88 της Συνθήκης Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τα Εθνικά Κοινοβούλια και το ευρωπαϊκού. Άρα δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα εθνικά, γιατί είναι από κοινού νομοθέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Εγώ είμαι υπέρμαχος του πρωταγωνιστικού ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μία μάλλον ένα από τα πιο ευάλωτα στοιχεία της λειτουργίας μας είναι η έλλειψη συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην αναζωογόνηση και επανικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, είσαμε μια κρίση την οποία πολύ καλά γνωρίζετε και δεν θα επαναλάβω. Ως προς τον αριθμό των μελών, εγώ δεν έχω κανένα θέμα μέσα στα πλαίσια της ε, διαπραγματευτικής εντολής. Απλώς ακούσαμε από πολλούς ότι θα πρέπει να είναι ένα ε, μικρό σχήμα για να είναι πιο ευέλικτο και πιο λειτουργικό. Και τέλος, και θα σταματήσω εδώ, θα ήθελα να πω το εξής. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες που σχετίζονται με δύο ζητήματα. Το ένα είναι γνωστό, που είναι το άρθρο 51. Στο άρθρο 51 που αναφέρεται στην τροπολογία μου 200 αφορά τις αρμοδιότητες αυτού του οργάνου ελέγχου. Και δεύτερον, ορισμένες άλλες ανησυχίες θα είναι απόρρια του κανονισμού, όπου θα οριστεί επακριβώς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και θα τελειώσω όπως άρχισα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τα οποία μου δώσαν πάρα πολλές γνώσεις και με βοηθούν στο έργο μου. Βασίζομαι σε σας και θα ήθελα να ξέρετε ότι και εγώ θα δείξω μεγάλη κατανόηση και ευελιξία προς τα δικά σας σχόλια. Συνάδελφοι, ένα μικρό σχόλιο από την Ανίτα Σάφερ και ο κύριος Μπον έχει στήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις διάφορες επικοδομητικές ε, συμβολές σας, για την κοινή ε, διοργάνωση αυτού του σώματος κοινοβουλευτικός ελέγχου, τη σημείωσα και εμείς θα στραφούμε ως ε, Γερμανική Βουλή με τα επιχείρηματά μας προς την Τρόικα. Συνοψίζω. Άκουσα διάφορους να λένε ότι πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να έχει σωστή γνώση και να ασκεί σωστά το δημοκρατικό έλεγχο. Την αποτελεσματικότητα θα την, επιτύχουμε, όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία, όχι μόνο μέσω των αριθμών των μελών, αλλά και μέσω του καθορισμού των κανόνων λειτουργίας. που είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Η αναγκαία ειδική γνώση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν σε αυτό το σώμα δεν συμμετέχουν μόνο οι δήμονες από τα κοινοβούλια, πρέπει να είναι μόνιμοι εκπρόσωποι, να υπάρχει συνέχεια στη δουλειά τους για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους. Είναι μια διαδικασία αυτό. Ο συγκεκριτής του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό της Europol τόνισε ότι αν θέλουμε να είναι κοινό όργανο ελέγχου και να λειτουργήσει, θα έχουμε δημοκρατικό έλεγχο της Europol. Και αν γίνει αυτό, και για να γίνει μάλλον αυτό, πρέπει να είναι δημοκρατικά οργανωμένος ο έλεγχος. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι ανανομισωτικό σώμα. Αυτό επιτρέπει να ε, αντιπροσωπευθεί ευρύτερα το φάσμα πολιτικών δυνάμεων. Αλλιώ δεν θα είναι δημοκρατικό έλεγχος. αλλιώς είναι. Α, για να είναι δημοκρατικό έλεγχο, χρειάζονται πάνω από μία συνεδρίαση το χρόνο, τουλάχιστον δύο. Και τώρα θα περιμένουμε ε, στην καινούργια, την καινούργια πρόταση της ε, Τρόικα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπον, ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ είχε θέσει ένα ερώτημα για εσάς. Μπορείτε να το απαντήσετε πολύ σύντομα, εφόσον έφυγε κιόλας προηγουμένως. Πρέπει να με συμβουλεύσετε τι συμβαίνει στι δικέ επιτροπέ όταν θέτει ένα μέλο μια ερώτηση και μεταφεύγει πριν ακούσει την απάντηση. Σίγουρα όλοι θα έχετε και από μια διαφορετική λύση. Στη δική μα περίπτωση σα αναγκάζουμε να απαντήσετε. Να του επιβάλλετε κυρώσει, προτείνω εγώ. Υπάρχουν πολλέ τέτοιε ε, μορφέ επιβολή πειθαρχία τι μέσα έχει το Ευρωκοινοβούλιο με μια έλλειψη κυρώσεων. Δύο είναι εδώ ε, οι λύσεις. Πρώτον, στενή συνεργασία με την Επιτροπή ε, Προπολογισμού και Ελέγχου του Προπολογισμού ε, του Ευρωκοινοβούλιο. Εάν θεωρείτε λοιπόν ότι η Europol δεν κάνει καλά τη δουλειά της ή θα πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της, σε κάποιον τομέα, μπορείτε να έρθετε ε, σε επαφή με αυτές τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όχι, δεν περίμενα πραγματικά <laughs> να μου απαντήσετε, ήταν ρητορικό. Δεύτερον, κατονομάζουμε μέσω του, των μέσων ε, ενημέρωσης. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόλ. Ήθελα πολύ συγκεκριμένα να ευχαριστήσω τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί ε, είναι πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα και αφαιρέσω το χρόνο για να έρθετε μέχρι εδώ. Θα έχετε δει ότι δεν ε, είναι πολύ πρόσφορο έδαφος για το, ένα γόνιμο διάλογο αυτές τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, γιατί δεν ε, μπορείτε να απαντήσετε και να δευτερολογήσετε κτλ. Όμως ε, όλα αυτά που αναφέρθηκαν σήμερα θα ληφθούν υπόψη στο σχέδιο πρότασης της Τρόικα και αυτό ήταν εξαιρετικά χρήσιμο εγχείρημα για μας. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστά αυτή η πρόταση γιατί εκτός από την Europol έχουμε μία σειρά νομοθετικών προτάσεων για το θεματολόγιο της ασφάλειας και ήθελα να το επισημάνω εδώ όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα ζητήματα τρομοκρατίας, ε, ξεπλήματος χρήματος κτλ, εθνικής κυριαρχίας ε, και ούτω καθεξής, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί από πλευρά κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γι' αυτό με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι ήρθατε τόσο πολύ εδώ και δώσατε πλήρη και σαφή εικόνα ε, των απόψεών σας για την πρόταση. Και ο κύριος Διαδεμέρα και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Είναι μεγάλο μας προνόμιο. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ευχαριστώ και ελπίζω να δοθεί και συνέχεια σε αυτή τη Σε Βέβαια η πρόταση ε, θα μας έρθει ε, τον Απρίλιο χάρη σας βοήθεια. Ευχαριστώ.